Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τώρα με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε ήδη μία μικρή καθυστέρηση και έχουμε μία λίγο φορτωμένη ημερήσια διάταξη γιατί κάποια σημεία της Πέμπτης έχουν συμπεριθεί στη σημερινή ε, διάταξη γιατί την Πέμπτη ορισμένοι συνάδελφοι ε, δεν μπόρεσαν ε, να παρουσιάσουν τα δικά τους θέματα. Βλέπετε όλοι ε, ποιες γλώσσες προβλέπονται εδώ. Η συνεδρίαση μπορεί να ακουστεί από το ίντερνετ. Και για τους περισσότερους που παρίστανται εδώ είναι πρόκειται κυρίως για μια επανάληψη. Στις 20 Απριλίου η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και μέσω του Επιτρόπου κ. Λεβαντόφσκι μας τον παρουσίασε σε μια συνεδρίαση και όλα τα κείμενα, όλα τα έγγραφα τα έχετε ήδη λάβει. Και ασφαλώς αργότερα όταν συζητήσουμε τον προπολογισμό του 2012 θα κάνουμε και τη σχετική συζήτηση. Ε, ήδη στα Κόμπου News έχουν ανακοινωθεί τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα ή όχι, λέει η Πρόεδρος. Έχει αναβληθεί ήδη το θέμα αυτό. Ωραία, λοιπόν. Έχει αναβληθεί το σημείο αυτό. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να έχουμε προβλήματα. Ούτε η κυρία Χολμάιερ ε, μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά δεν μπορεί να έρθει ούτε την Πέμπτη. Άρα λοιπόν, ε, όσον αφορά την πολιτική των ε, κτηρίων, θα το διαγράψουμε από την ημερήσια διάταξη και θα αναβάλουμε το σημείο αυτό για την προσεχή συνεδρίαση. Και μένα η δική μου γνωμοδότηση, οι δικέ μου προτάσεις γνωμοδότησης για την ΕΝΙΖΑ και την ΕΜΖΑ, η οποία έχει περισσότερα καθήκοντα, η ΕΜΖΑ, και η ΕΝΙΖΑ, η οποία θα πρέπει να έχει μια καινούργια νομική βάση και θα πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα γιατί ναι μεν θα είμαι εγώ παρούσα και την πέμπτη αλλά δεν ξέρω ε, πότε θα πρέπει να πάω στη διάσκεψη των ε, Προέδρων για να παρουσιάσω την πρόοδο των εργασιών και την έκθεση ΣΟΥΡ. Ε, γι' αυτό είναι καλύτερο να το κάνουμε ήδη σήμερα. Και έτσι θα έχω το ελεύθερο να εγκαταλείψω την έσοδα φύγω όταν χρειαστεί. Άρα λοιπόν θα κάνουμε τη συζήτηση σήμερα. Ξέρετε ότι έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα για την ε, κατάθεση των τροπολογιών. Τώρα, όσον αφορά την ε, σειρά των θεμάτων που σας πρότεινα στον, ε, που, που βρίσκω στον αδεικτικό μου κατάλογο, Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά. 1, 2, 3, τα ολοκληρώσαμε. 7, 6, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 και 13. Άρα λοιπόν, ε, θα ανακατέψαμε λίγο και θα ξεκινήσαμε με το 7 που πρόκειται για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και θα ήθελα να παρακαλέσω την Μπάρμπαρα Ματέρα να μας κάνει μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω μια νέα αίτηση για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση από το κράτος του Βελγίου σκοπός είναι να στηρίξουμε τους εργαζομένους της πολυεθνικής, της αμερικανικής ε, πολυεθνικής που ενεργεί στην αυτοκινητοβιομηχανία, την General Motors. Υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος από την οικονομική κρίση και έχει μειωθεί η δυνατότητα η αγοραστική των ε, καταναλωτών. Οπότε ε, η ζήτηση και για παραγωγή οχημάτων. Άρα η General Motors αναγκάστηκε να πωλήσει 2.834 εργαζομένους και της πολυεθνικής και των θεκατρικών των εργοστασίων της που πολλούν σιλιανική. Τώρα, το βελγικό κράτος και μετά από συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους ζητά χρηματοδότηση από το ΦΕΑΓ για ένα ποσό των 9.600.000 ευρώ περίπου. Εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα αίτημα που προέρχεται από πολυεθνική. Και θέλω να θυμίσω τι συνέβη τον περασμένο μήνα όταν υπέβαλα το αίτημα της Unilever και άλλη μια πολυεθνική. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι από τους σοσιαλιστές υποβλήθηκε τροπολογία η οποία εγκρίθηκε στην Ολομέλεια με 135 ψήφους υπέρ και 280 κατά. Αλλά αυτό μας ε, είχε δημιουργήσει πολλούς ενδιασμούς, διότι αυτό, αυτή η τροπολογία θα παρά την υπερβολικά τους χρόνους κινητοποίησης των απαιτούμενων ποσών, όχι υπέρ της Unilever ούτως ή άλλως, αλλά για τους εργαζομένους της Unilever που είχαν απολύθει γι' αυτό. Λοιπόν, για την General Motors έχω συμπεριλάβει την παράγραφο 6. Παράγραφο 6 που σήμερα ήθελα όλοι σας να την ε, κοιτάξετε διότι λέει ότι θεωρεί το ζήτημα των πολυεθικών ε, εταιριών που αναδιαρθρώνονται ή μετατοπίζονται προκαλεί απολύσεις. Οπότε η παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να λυθεί υπόψη στην επόμενη αναθεώρηση του πλαισίου εντός του πιλητού και το τομείο αυτό, ώστε να μην δυσκολεύεται η πρόσβαση των εργαζομένων στα κονδύλια του Ταμείου. Ελπίζω ότι μπόρεσα εδώ να καλύψω τις ανησυχίες κάποιων συναδέλφων που ούτω ή άλλω μπορεί να καλύπτεται και από μια παράγραφο έτσι με πιο ήπια διατύπωση από ότι η τροπολογία που είχαν υποβάλει προηγουμένω οι σοσιαλιστέ. Να θυμόμαστε πάνω απ' όλα ότι το ταμείο αυτό δεν είναι ένα ταμείο που ωφελεί τι εταιρείε, τι πολυεθνικέ. Είναι ένα ταμείο που αφορά τα άτομα. Πηγαίνει απευθεία και απευθύνεται απευθεία στου εργαζομένου. Να θυμίσω ότι προβλέπεται συγχρηματοδότηση από το κράτο, ιδίω ό,τι αφορά το έλεγχο έτσι ώστε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες απόλυσης μέσω των συλλογικών συμβάσεων και βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις ε, συλλογικές απολύσεις. Και την εθνική νομοθεσία. Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι δεν πιστεύω ότι οι πολυεθνικές ή οι επιχειρήσεις ε, επιλέγουν να απολύσουν σε ενός εργοστασίου περισσότερο εις βάρος των εργαζομένων κάποιου άλλου ή υπέρ Και σε κάθε περίπτωση Να πω ότι η υποβολή τροπολογιών, όπως αυτή που υποβλήθηκε από τους σοσιαλιστές, με αφορμή την προηγούμενη έκθεσή μου για τη Unilever, ουσιαστικά παρατείνει τους χρόνους εκταμίευσης των ποσών υπέρ των εργαζομένων. Σας παρακαλώ λοιπόν, εάν πιστεύετε ότι εδώ θα ωφεληθούν οι πολυεθνικές. Παρακαλώ να βγείτε από αυτή την πλάνη. Εδώ μιλάμε για εργαζομένους. Ε, μπορεί να είναι εργαζόμενοι πολυεθνικών, αλλά δεν πάβουν να είναι εργαζόμενοι. Ελπίζω ότι υπήρξα σαφής, διότι πραγματικά μου φάνηκε άστοχη η τροπολογία που έχει υποβληθεί από τους σοσιαλιστές. Να θυμίσω τις ημερομηνίες για την υποβολή τροπολογιών για αυτή τη νέα έκθεση. Η προθεσμία λέγει στις 11 Μαΐου και η έκθεση αυτή θα ψηφιστεί στις 23 ή 24 στην Επιτροπή Προπολογισμών και θα πάει στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω ότι δεν ήμουν ε, πολύ γρήγορη. Ευχαριστούμε πολύ. Η γερμανική διερμηνία ε, τα κατάφερε. Άρα δεν ήταν μεγάλη ταχύτητα, τουλάχιστον με τη γερμανική ε, διερμηνία. Ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ε, και ε, σε σχέση με το νόημα του ταμείου αυτού θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους και όχι την εργοδοσία. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ε, υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στην εισηγήτρια. Σαφώς είμαι υπέρ του να μπορούμε να εκταμιεύσουμε τους απαραίτητους πόρους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την General Motors. Έχω όμως και ένα ερώτημα. Εργαζόμαστε κυρίω με την εκταμείευση των πόρων αυτών για, για του εργαζομένου των επιχειρήσεων αυτών. Η κυρία Ματέρα αναφέρθηκε όμω και σε μια τροπολογία των σοσιαλιστών, καθώ επίση και σε μια τροπολογία την οποία θα αναδιατύπωνε προκειμένου να μπορέσουν τα χρήματα να φτάσουν πολύ πιο γρήγορα στους εργαζομένους. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το ακόλουθο. Συζητάμε αυτή τη στιγμή μόνο την αποστολή των πόρων αυτών προ την General Motors τη Αμβέρσα ή θέλουμε μέσω της τροπολογίας αυτής να πλουστεύσουμε λίγο την όλη διαδικασία εκταμίευσης των πόρων προκειμένου αυτά να φτάνουν πιο γρήγορα στους αποδέκτες τους. Μιλάμε λοιπόν μόνο για την General Motors σε σχέση με αυτή την τροπολογία ή γενικότερα για την ακολουθητή διαδικασία. Μπάρμπαρα. Μιλούσα για μια τροπολογία που είχαν υποβάλει οι σοσιαλιστές ως ομάδα, όπου ζητούσαν μεγαλύτερη σαφήνεια για τον τρόπο κατά τον οποίο ορίζεται ο παραλήπτης των ε, πόρων ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τις πολυεθνικές. Ζητούσαν να επαληθεύεται η δημοσιονομική κατάσταση, η φοροδιαφυγή και τι βοήθειες δίνουν τα κράτη που, στις οποίες βρίσκονταν και είχαν την έδρα τους οι πολυεθνικές. Δηλαδή ζητεί το από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνεται περισσότερος έλεγχος. Όπως είπα και προηγουμένως, οι έλεγχοι γίνονται ούτως ή άλλως εκ των προτέρων. Εφόσον θεωρούμε ότι υπάρχει συγχρηματοδότηση 35% από το κράτος μέλος, επί το οποίο εδράζεται μια πολυεθνική. Εάν δεν υπάρχει σαφήνεια, δεν πρόκειται να διαθέσει πόρους ούτως ή άλλως το κάθε κράτος. Θεωρείται δεδομένο. Ähm, Αν το κατάλαβα καλά, λέει η Μπάρμπαρα Ματέρα ότι η παράγραφος 6 το συμπεριλαμβάνει αυτό με κάπως πιο ήπια διατύπωση, πιο αποδυναμωμένη μορφή. Μάρτα Ανδρέασαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητήσαμε το ζήτημα της κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από το γεγονός ότι ε, δεν προβλέπονται απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όντως το Ταμείο αυτό χρησιμοποιείται για την ε, επανακατάρτιση των ε, εργαζομένων αυτών που έχουν απολυθεί από διάφορες εταιρείες. Το Ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για την ε, κατάρτιση των εργαζομένων σε ένα συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο. Βλέπουμε όμω ότι ο συγκεκριμένο τομέα που συζητάμε τώρα, η αυτοκινητοβιομηχανία, είναι ένα τομέα που εξαφανίζεται. Σε ποιο κλάδο πρόκειται να ε, καταρτήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Θα γίνουν ειδικοί σε θέματα πληροφορικής ή σε κάτι άλλο. Γιατί νομίζω ότι όλη η σε κατι αλλο γιατι νομιζω οτι ολη χρηση του ταμείου αυτού αυτή τη στιγμή τίθεται ένα αμφιβόλο. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Αναφερόμαστε τώρα στη General Motors και λέμε ότι έχει διάφορα προβλήματα λόγω της κρίσης. Δεν λέμε όμως ότι ενδεχομένως η General Motors να έχει προβλήματα στο Βέλγιο επειδή άνοιξε εδώ η αγορά στους Ασιάτες κατασκευαστές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει συμφωνίες εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες αυτές που ουσιαστικά έχουμε διευκολύνει τις συνθήκες για τις ασιατικές εταιρείες. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει σε σχέση με το ταμείο αυτό να σταματήσουμε λίγο και να σκεφτούμε αν πραγματικά χρησιμοποιείται σωστά και αν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Ευχαριστώ. Ναι, ασφαλώς αληθεύουν όλα αυτά. Μόνο που αυτή τη στιγμή εδώ είναι το λάθος σημείο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν συζητούμε δηλαδή το Ταμείο προσαρμογή στο σύνολό του, αλλά συζητούμε κατά πόσο αυτό το οποίο αποφάσισε θετικά η Επιτροπή ανταποκρίνεται στο αίτημα του Βελγίου όσον αφορά τα, την εκταμίευση κονδυλίων από το Ταμείο Προσαρμογής. Η Κομισιόν είπε ότι πληρούνται όλε οι προποθέσει οι οποίε ε, πρέπει να πληρούνται κατά την υποβολή ενός τέτοιου αιτήματος. Και εμεί θα πρέπει να αποφανθούμε σχετικά, όχι μόνο εμεί βεβαίω, αλλά εμεί, μέσω τη δική μα γνωμοδότηση και η Επιτροπή απασχόληση μέσω τη δική τη έκθεση, θα πρέπει να αποφανθεί κατά πόσο έχει δίκιο η Επιτροπή, η Κομισιόν ή όχι. Ε, παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι το να εξτάσουμε εδώ να συζητήσουμε εμπορικέ συμφωνίε. Υπάρχουν άλλες δύο παρεμβάσεις και στη συνέχεια θα κλείσουμε αυτό το σημείο. Όποιος επιθυμεί να καταθέσει κάποιες τροπολογίες ε, μπορεί να το πράξει μέχρι τις 11 Μαΐου. Ιζαμπέλ, θέλεις να πάρεις το λόγο? Όχι, ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο συντομία κυρία Πρόεδρε, χωρίς να θέσω να αμφιβόλω την ε, ύπαρξη του Ταμείου και την υποστήριξη της ε, κατάρτισης των απολυθέντων εργαζομένων. Φυσικά εγώ υποστηρίζω αυτή την ιδέα, αλλά θα ήθελα να πω ότι ε, ποτέ δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή τόσα οχήματα στον κόσμο, ούτε τόσα χρήματα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αντίθετα όσα λέγονται. Δεύτερον, είναι πέντε δις ο τζίρος της εταιρείας. Ε, άρα λοιπόν, ε, κατά πάσα πιθανότητα εμεί ε, δίνουμε χρήματα, αλλά για την τελή υπόθεση. Αλλά είναι κάπως σοκαριστικό να διαπιστώνουμε ότι μια βιομηχανία που έχει τόσα κέρδη, ε, προχωρά σε μια τέτοια πώληση εργαζομένων. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ε, ξέρουμε τι θέλουμε να, τι θα πρέπει να ψηφίσουμε στη συνέχεια και ακούσαμε και την πρόταση της Μπάρμπαρα Ματέρα για την έκθεση αυτή. Η Μπάρμπαρα έχει πάλι το λόγο. Πρόεδρε, πολύ γρήγορα για να κλείσουμε. Ε, επειδή βλέπω ότι η συζήτηση για αυτό το ταμείο και για τη χρήση του ενδιαφέρει πάρα πολύ τους συναδέλφου, θεωρώ ότι καλό θα ήταν σε πρώτη φάση να στηρίξουμε αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε εδώ, γιατί υποβάλλω και ένα ερώτημα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στην επόμενη Ολομέλεια να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Του περασμένου μήνε, λόγω των ε, ανηλυμένων δεσμεύσεων των ΜΕΝ και των ΔΕ, δεν μπόρεσαμε να το συζητήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια συζήτηση επί τη ουσία για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια και ζητώ τη στήριξη όλων των συναδέλφων για να συμβεί αυτό. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν, αλλά θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι δεν έχει περάσει πολλές καιρός από τότε που καταρτήσαμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Υπεύθυνος για αυτήν ήταν ο συνάδελφος κ. Πόρτας και ήταν πραγματικά μια ιδιαίτερως ε, περιεκτική έκθεση. Ωραία. Κλείνουμε εδώ αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ένα σημείο που ασφαλώς είναι, ιδιαίτερος, είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που δεν είναι και τόσο δημοφιλές θα έλεγα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το δημοσιονομικό κανονισμό και η Ίγκε Γκρέσλε ως συνήθως θα κάνει μια παρουσίαση. Αλλά θα ήθελα να πω σε όλους τους ε, συναδέλφους ότι οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχουν προσκληθεί στη δική μας συνεδρίαση εάν έχουμε τη δυνατότητα με αυτούς από κοινού να συζητήσουμε το θέμα αυτό και την Πέμπτη οι συντονιστές να συζητήσουν για το νέο χρονοδιάγραμμα και να αποφασίσουν κατά πόσο αυτό το νέο πρωταθέν χρονοδιάγραμμα είναι εντάξει. Ε, Λοιπόν, τώρα η Ίγκεμπορκ θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Θα, ε, θα είμαι αρκετά σύντομη. Με προσκάλεσα να αναφερθώ σε κάποια βασικά θέματα και εδώ το θέμα είναι πάλι επιδοτήσει και οι μεταφορέ των πιστώσεων. Μεταφορέ γιατί μια αρμοδιότητα αυτή τη Επιτροπή ε, είναι αυτή. Και επειδή πάρα πολλέ τροπολογίε αναφέρονται στο θέμα αυτό των μεταφορών. Ε, εν τω μεταξύ έχουμε την ε, έκθεση στα αγγλικά. Δεν ήταν ε, πολύ εύκολο να προσλάβει την οριστική τεχνική τη μορφή γιατί υπάρχει ένα νέο σύστημα εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τη Γραμματεία γιατί ξέρω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνουν κάποιες ε, τεχνικές ε, αλλαγές. Αρχικά ήταν 100 τροπολογίες και πλέον είναι 200. Ε, ε, τώρα με το νέο σύστημα πρέπει να ασχοληθεί κανείς με την κάθε χωριστή παράγραφο. Εγώ έκανα 100 τροπολογίες και ε, ε λυπούμε ε, για αυτή την ε, κατάσταση, αλλά δεν ήταν δυνατόν να συνοψιστούν περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά τι μεταφορέ, τα transfers, η έκθεση υπάρχει στα αγγλικά και αν υπάρχουν κάποιε ασάφειε, παρακαλώ να έρθει σε επαφή μαζί μου και πραγματικά είμαι ευγνώμων προς τον καθένα ο οποίος είναι διατεθειμένος να διαβάσει την έκθεση. Έχουμε τα παλιά άρθρα 23 και 24 του κανονισμού στο πλαίσιο του προπολογισμού του 2011 έχουν γίνει κάποιες μεταβατικές συμφωνίες που θέλουν να εντάξουν τη συνθήκη της Λισαβόνα στο δημοσιονομικό κανονισμό. Γι' αυτό οι βασικές αλλαγές για αυτές τις μεταβατικές συμφωνίες αφορούν την διαγραφή των υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών πληρωμών. Αλλά η Επιτροπή πλέον έκανε κάποιες αλλαγές εδώ ε, στον δημοσιονομικό κατανομισμό και μας ε, προτείνει τα, ε, μας προτείνει κάτι που αφορά τις μη υποχρεωτικέ δαπάνες. Δηλαδή αυτό το οποίο ισχύει για τις μη υποχρεωτικέ δαπάνες τώρα θα πρέπει να ισχύει και τις υποχρεωτικέ δαπάνες και για παράδειγμα έχει προβλέπει 100 εκατομμύρια πληρωμών, υποχρεώσεων πληρωμών ε, και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό καθώς και η προθεσμία που προβλέπει για τις τρεις εβδομάδες. Δηλαδή προτείνει κάποιες αλλαγές η Επιτροπή που πραγματικά συρρυκνώνουν τα δικαιώματά μας και τις αρμοδιότητες και αυτό δεν το αποδέχτηκα. Γι' αυτό έχουμε τις τροπολογίες 22 έως 30 έως 33 συγγνώμη, που έχουν σαν σκοπό να αποκαταστήσουν την προηγούμενη κατάσταση όσον αφορά τις μη υποχρεωτικές δαπάνες. Και υπάρχει και μια πολύ καλή σημείωση της γραμματείας που θα ήθελα να την κοινοποιήσω προς όλους όσου επιθυμούν να μάθουν κάποια πράγματα παραπάνω. Το ελεγκτικό συνέδριο, στη δική του γνωμοδότηση για τον δημοσιονομικό κανονισμό, επισημαίνει επίση ότι αν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συντόμευση από έξι εβδομάδες σε τρεις εβδομάδες όσον αφορά τις προθεσμίες θα έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ πραγματικά έχουμε πάρα πολύ, πολλά καλά επιχειρήματα στο δικό μας πλευρό για να μην ακολουθήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 22-33 τροπολογίες οδηγούν στην διατήρηση της προηγούμενης κατάστασης όσον αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τις... Ε, ε, το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και οι συγκητές έκαναν πολλές συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους και από τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κάναμε ένα στρογγυλό τραπέζι. Είχαμε την έκθεση Καβάλιο, της Ήτρε, την οποία εμείς επηρεάσαμε και είχαμε πολλούς γύρους συζητήσεων, ακόμα και με τους διαφόρους μάνατζερ και έχουμε και την ε, αναπτύξη ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία προσπαθεί να κάνει μια απλούστευση των δικών μας τροπολογιών. Ε, οι δικές μας τροπολογίε εν μέρη είναι αποτέλεσμα της συζήτησης με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς και έχουν τον εξή σκοπό οι δικές μας τροπολογίε Θέλουμε μία απλούστευση για επιτάχυνση των διαδικασιών. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις μεταξύ κανονισμού, εκτελεστικών διατάξεων και οδηγιών που δίδονται στους ε, δικαιούχους. Ε, ο κανονισμός, υπάρχουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, οι συνθήκες και ο τομεακός ε, κανονισμός. Έχουμε έξι διαφορετικά νομικά κείμενα και αυτά τα έξι διαφορετικά νομικά κείμενα θέλουμε να τα αντικαταστήσουμε με έναν ξεκάθαρο νομικό κανονισμό. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ξεπεράσουμε τις ενδεχόμενες αντιφάσεις μεταξύ αυτών των νομικών κειμένων. Επίσης όσον αφορά ε, την εφαρμογή του άρθρου 390 τις της ε, ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, αυτό δεν αφορά καθόλου ζητήματα μικροδιαχείρισης, αλλά πρόκειται για την εφαρμογή της συνθήκης τη Λισαβόνας και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έκανε κάποιες προτάσεις σε σχέση με τα τμήματα των εκτελεστικών διατάξεων, τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ίδιο τον κανονισμό. Υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις αποστήλαμε στις ομάδες εργασίε και ε, εδώ δεν πρόκειται για μυστικές ε, διαδικασίες, αλλά πρόκειται για την ε, συμπερίληψη διαφόρων τμήματων τα οποία έχει προτείνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μικρές επιδοτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ, μέχρι 50.000 ευρώ το ορίζουμε μέσω του ποσού. Και είπαμε ότι όσο μικρότερο, μικρότερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο είναι το διοικητικό άχθος. Και αυτό θα πρέπει να πηγαίνει μέχρι την αποδοχή του αιτήματο. Πρόκειται για υδροπολογία υπερθών 135 που φορά αυτές τις μικρές επιδοτήσεις. Ε, μετά έχουμε τροπολογία 138 που πρόκειται για τα σταθερά ποσά, τα lump sums, ε, το flat rate financing. Όταν ορίζονται τέτοια ποσά, δεν θα πρέπει να υπολογίζονται άλλη μια φορά εκ των υστέρων ε, και έχουμε, γιατί με τον τρόπο αυτό καταργείται η επλούστευση που επιθυμούμε και γνωρίζουμε ότι ε, θα υπάρξουν ίσως κάποια προβλήματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ ξεκάθαρος κανονισμός. Επίσης ασχοληθήκαμε με την τροπολογία 138 που αφορά τα ποσά κάτω από 5.000 ευρώ θα πρέπει οι δικαιούχοι να μην ε, αποδεικνύουν ε, τις δαπάνες τους σε σχέση με, τα, με την απορρόφηση αυτών των ποσών. Ε, υπάρχει αύξηση των σταθερών ποσών και θεωρώ αυτό είναι σημαντικό. Στη συνέχεια έχουμε τα επιλέξιμα, το επιλέξιμο, τα επιλέξιμα κόστη αυτοί οι καθορισμοί μέχρι στιγμής ήταν ιδιαίτερως αντιφατικοί. Έχουμε, για παράδειγμα, την, ε, τον, το ζήτημα του φόρου, ο οποίος θα πρέπει να υπολογίζεται, επίσης τις διοικητικές δαπάνες για το λειτουργικό κόστος των ε, μη κυβερνητικών οργανωσμών ε, και υπάρχει εδώ μια αύξηση της τάξης του 10% για τα ποσά που δεν υπερβαίνουν τις 250.000 ε, ευρώ. Και η τροπολογία 143, η οποία αφορά την ε, συγχρηματοδότηση in kind, Και εδώ προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τα μικρά ποσά κάτω από 5.000 ευρώ όπου ε, δεν είναι δυνατόν, ε, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται, δεν χρειάζεται μια αιτιολόγηση για την απόρριψη αυτών των ποσών. Έχουμε έναν κανόνα στο δημοσιονομικό ε, κανονισμό, έχουν κανόνα στο δημοσιονομικό κανονισμό που μέχρι στιγμή ε, δεν έχουν εφαρμοστεί και δημιουργούν πολλά εμπόδια και γι' αυτό προσπαθήσαμε να του διαγράψουμε. Έχουμε επίση ε, την τροπολογία 148 που δεν ενθουσιάζει καθόλου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τη διαδικασία υποβολή αιτήσεων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μετά από έξι ομα... ε... μήνε. Επίσης το ζήτημα των εγγύσεων, την ε, τροπολογία υπαριθμών 152 και επιθυμούμε να γίνει μια ανάλυση του κινδύνου για ποσά κάτω από 5.000 ευρώ, για πολύ μικρές επιδοτήσεις, θέλουμε εδώ να μην απαιτούνται πλέον εγγύσεις για τα ποσά αυτό. Και αυτό θα βοηθήσει, θεωρούμε, πολλούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς στον τρίτο κόσμο. Επίσης, έχουμε την ε, τροπολογία 148, ε, που αφορά πάλι τις ε, προθεσμίες ε, μεταξύ 3 και 10 ετών, η πρώτη τριβολογία 158, εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ρύθμιση με το ελεγκτικό συνέδριο και όσον αφορά το κλείσιμο των λογαριασμών, πρόκειται για το διάστημα για το κλείσιμο των λογαριασμών. Και θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια επιτάχυνση κάποιων διαδικασιών. 159-160 που αφορά τις επιτροπές clearing μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης και οι οποίες θα ασχοληθούν με την ενή ερμηνεία μεταξύ των κανόνων από τις διάφορες ε, γενικές ε, ε, διευθύνσεις. Οι 174 αφορά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Επίσης έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και βλέπουμε ότι μέσω των τεχνικών προβλημάτων αυτή τη στιγμή έχουμε προγραμματίσει τον Ιούλιο να κάνουμε μια κοινή ψηφοφορία μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια να γίνει η, οριστική ε, η τελική ψηφοφορία. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα, χιλιάδες άλλα θέματα τα οποία είναι πολύ πιο σεξι και πολύ πιο ενδιαφέροντα αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα θέματα γιατί αλλιώς θα μας πέσουν στο κεφάλι τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε το σθένος, να αλλάξουμε κάποια πράγματα όπως οφείλουμε να το πράξουμε και θα πρέπει να κρατήσουμε εμείς τα νήματα στα χέρια μας για τις αλλαγές αυτές. Όσον αφορά τις ε, μεταφορές ε, πιστώσεων, ε, πάντοτε βρισκόμαστε στην αντιπαράθεση με το Συμβούλιο για τα θέματα των πληρωμών και μέχρι στιγμής ε, πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να κάνουμε πολλές υποχωρήσεις. Γι' αυτό έκανα αυτές τις ε, προτάσεις για τις ε, αλλαγές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι όταν μας κάνει μία παρουσίαση και σε ακούμε και εμείς προσεκτικά, τα πράγματα ξεκαθαρίζονται πολύ περισσότερο. Λοιπόν, η Μαρία Καβάλιο, ο κύριος Οντί, Μάνκα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να <clears throat> ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για το πολύ σημαντικό έργο και το ανοιχτό πνεύμα που επέδειξε, συνεργαζόμενοι με τα μέλη και της ε, Ήτρε. Προσπαθήσαμε με την έκθεση αυτή να πλουστεύσουμε τους κανόνες για τη συμμετοχή στα προγράμματα ανάπτυξης και καινοτομίας με βάση κάποιες συστάσεις. Συστάσεις που εγκρίνουν και προτρίνουν κανονισμούς, ε, αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό οι ουσιαστικές συστάσεις που ζητούν αλλαγή ακριβώς εκεί επέμεναν στις αλλαγές ε, τροποποιήσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην οδό της απλούστευσης και είναι ζωτική σημασία να το κάνουμε το βήμα αυτό και στην κατεύθυνση που τώρα ακολουθούμε. Χάρη λοιπόν Χάρη λοιπόν στην αποδοχή των ε, εγκεκριμένων πρακτικών για τα λογιστικά πρότυπα, την απλούστευση των, του, της καταγραφής χρόνων και προθεσμιών, των κριτηρίων προχρηματοδότησης, της χρήσης κατά αποκοπήν ποσών, την μείωση ανάγκης για ελέγχους εκ των υστέρων και υπερβολικές διορθώσεις και τέλος, τον διάκριση διαδικασιών, της όλης μάλλον διαδικασίας, του κύκλου των προγραμμάτων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για όλους τους ενδιαφερομένους που υποβάλλουν αιτήσει για χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω ξανά την εισηγήτρια που δέχτηκε τις δικές μας απόψεις και συνεργάστηκε τόσο στενά με τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσει των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ερευνητών καλύπτονται και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Ευχαριστώ. Ähm, ευχαριστώ πολύ, κύριο Σοντή. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που προσκαλέσατε μέλη από τις άλλες επιτροπές για τη συζήτηση αυτή που κάνετε για, την, ε, για το δημοσιονομικό κανονισμό. Θα ήθελα να σε τρία στοιχεία, κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχει έρθει η στιγμή αυτή που θα πρέπει να δημιουργήσουμε στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Βλέπουμε όλο και περισσότερο, σε εξελίσσει Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι χρειάζεται να κάνουμε όλο και περισσότερες επενδύσεις οι οποίες είναι πολυετής και ιδιαίτερα σημαντικές. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, ο το τρέχον σύστημα προπολογισμού, κατάρτιση προπολογισμού δεν ευνοεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να αναφερθώ για παράδειγμα στο Ήτερ ή στον Καλιλαίο, όπου χρειάστηκε να κάνουμε πολύ σημαντικέ επενδύσει. Δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για επενδύσει στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση να πω ότι οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή ε, με φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Δεν καταλαβαίνω πώ θα εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο φορολογούμενο ότι αποδεχόμαστε επίπεδα κινδύνου ούτε ενεχόμαστε πολύ ψηλά επίπεδα κινδύνου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει περαιτέρω συζήτηση για το ζήτημα αυτό. Και τέλος, δύο ακόμα παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά τις προθεσμίες για τον έλεγχο του προπολογισμού και για την απαλλαγή. Είμαι μέλο Επιτροπής Ελέγχου των Προπολογισμών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει αυτό το μήνα την απαλλαγή για το 2009. Νομίζω λοιπόν ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι ιδιαίτερα μακρά και εκτενή και όσο και να είναι πολύπλοκος ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό, θα πρέπει να προβλέπετε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο να είναι πολύ πιο γρήγορο. Εμείς αυτή τη στιγμή ψηφίζουμε την απαλλαγή πάντα δύο χρόνια μετά το κλείσιμο των λογαριασμών. Προτείνω λοιπόν η διαδικασία αυτή να επιταχυνθεί. Το ελεκτικό συνέδριο να ολοκληρώνει εργασία του και αυτό γρηγορότερα. Άλλωστε, το ελεκτικό συνέδριο ελέγχει του λογαριασμού πάντα κάθε έτο σε τήσια βάση. Μέχρι τι 30 Ιουνίου, λοιπόν, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προθεσμία αυτή μετά το κλείσιμο των λογαριασμών και στη συνέχεια εμεί να παρεμβαίνουμε το δεύτερο εξάμεινο του έτου που έπεται του κλείσιμου των λογαριασμών. Δηλαδή, πριν τις 30 Ιανουαρίου από το ακόλουθο έτος. Επίσης, στη μεταρρύθμιση αυτή δεν αναφερόμαστε πολύ στην καταπολέμηση της απάτης. Η κατάσταση βελτιώθηκε όσον αφορά τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των παρατυπιών και των σφαλμάτων. Υπάρχουν όλο και λιγότερα σφάλματα, αλλά γίνονται όλο και περισσότερες απάτες. Και ορισμένοι ελεκτές θεωρούν ότι όσο ελέγχουμε περισσότερο τα σφάλμα και τις παρατυπίες τόσο θα καταπολεμήσουμε περισσότερο και την απάτη. Δεν ισχύει πιστεύω κάτι τέτοιο γιατί οι απαταιώνες έχουν τεχνικές που διαφεύγουν του ελέγχου των λαθών, των σφαλμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι στον κανονισμό αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή παράγραφος για την καπολέμηση της απάτης. Μπορούμε στη τελευταία ανάλυση να ανεχτούμε κάποια σφάλματα αλλά δεν μπορούμε να ανεχτούμε καμία απάτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βλαντιμίρ Μάνκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ δύσκολη αυτή εργασία την οποία έκανε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία τροπολογία που έχει να κάνει με την πολιτική και τα κτίρια για τη μεταφορά χρημάτων, πόρων όσον αφορά την πολιτική κτηρίων. Προβλέπετε εδώ πέρα ότι θα γίνουν κάποιες μεταφορές πόρων και είναι δυνατόν να γίνουν για το επόμενο χρηματοοικονομικό έτο, δημοσιονομικό έτο. Αυτό δεν συνάδει όμω με την πολιτική που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή για τα κτίρια, ούτε συνάδει με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να θέσω σε σχέση με αυτό κάποια ερωτήματα. Δεν ξέρω αν ο συντάκτη των τροπολογιών αυτών, η κυρία Μόνικα Ρωμαέλη, θα μπορούσε να απαντήσει σε ερωτήσει αυτέ, Θα ήθελα πάντω να γνωρίζω ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία στηρίζουν μια τέτοια δυνατότητα και δεύτερον, για ποιο λόγο ο συντάκτης των τροπολογιών απαιτεί ειδικά να ισχύουν οι διατάξεις αυτές για την πολιτική κτηρίων και γιατί όχι και στις υπόλοιπες πολιτικές. Και τέλος, ποιε ήταν οι επιπτώσει των προτάσεων αυτών, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μιλάμε για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κτίρια τα οποία έχετε κατά νου για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση που αφορά τις μεταφορές. Νομίζω ότι συμφωνώ με Ίγκε στο ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνουν πολύ μακριά υπερβολικά μακριά. Από την άλλη, το σύστημα όσο έχει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως αντιμετωπίζουμε αυτές τις μεταφορές αυτή τη στιγμή, επιδέχεται το σύστημα κάποιων βελτιώσεων. Στην ομάδα μας η συζήτηση πηγαίνει προς την ε, κατεύθυνση όχι κατά ανάγκη μιας αποκατάστασης της προηγούμενης ε, κατάστασης, αλλά ε, στο να προβληματιστούμε σε σχέση με μία μοιρασιά σε τρία κομμάτια, σε τρεις άξονες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής εάν έχουμε κάποια στοιχεία εν σχέση με το μέσο όρο των μεταφορών πιστώσεων. Γιατί ποσά μιλάμε ανά έτος προπολογισμού. Γιατί στη συζήτησή μας ε, ε, θεωρούμε ως προϋπόθεση ότι οι μικρές μεταφορές δεν είναι προβληματικές. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή να εξασφαλίσουμε έναν ευέλικτο προϋπολογισμό μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό εφόσον βεβαίως ενημερώνεται προηγουμένως η Επιτροπή. Για ένα δεύτερο τμήμα μεταφορών επιθυμούμε να προηγηθεί μια γνωμοδότηση. Δηλαδή η Επιτροπή Προπολογισμού να προβεί σε μια αξιολόγηση του κατά πόσο ε, θέλει να συζητήσει μια μεταφορά πιστώσεων και εφόσον το κάνει να την εγκρίνει. Και υπάρχει και μια τρία κατηγορία ε, μεταφορών πιστώσεων κάτω από τα πρωταθέντα κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι ε, χαμηλότερο το ποσό από τα 5.000 ευρώ. Ε, Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πάνε υπερβολικά μακριά και των προβληματισμών των σκέψεων τη γκε. Δηλαδή, ε, κατ' ουσία, να εμείνουμε ε, στι προηγούμενε διαδικασίε, διαδικασίες, διαδικασίε, ε, και σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις ε, ίσως εκεί να σκεφτούμε κάποια αλλαγή. Αυτή την πρόταση θα ήθελα εγώ να υποβάλω προς συζήτηση. Ναι, ε, καταρχήν θα συγκεντρώσουμε όλες τις απόψεις. Ο Λάσλο Σούριαν έχει το λόγο. ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις ε, επενδύσεις ακούσαμε από την ε, Κοκομπού ότι θα, θα ήταν, αναγκαία, να υπάρξει μια γραμμή του προϋπολογισμού όταν ε, το ζητούμενο είναι να ξεβρεθούν τα κονδύλια για κάποιο πρόγραμμα σε ένα έτος προπολογισμού, δυσκολευόμαστε όταν για παράδειγμα ε, στον Καλλιλέο δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη θέση, δεν προβλέπεται κάποια γραμμή του προπολογισμού για παράδειγμα για το πρόγραμμα Καλλιλέο. Και ένα άλλο θέμα. Ίσως το Συμβούλιο θα έπρεπε κάποτε να έχει τη δυνατότητα να ορίζει ένα ποσό κατά αποκοπήν. Και ίσως ε, παρόλο που ε, έχουμε προχωρήσει ίσως υπερβολικά μακριά στην έκθεσή μας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ίσως θα έπρεπε να έχουμε δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, θέλει να έχει μια μακροπρόθεσμη πολιτική κτηρίων θα πρέπει να μεριμνήσει για περισσότερη διαφάνεια αντί για τις ισχύες της διαδικασίας, δηλαδή να προσπαθεί κανείς να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα κονδύλια από εδώ και από εκεί. Και όσον αφορά τις μεταφορές, εδώ πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει να υπάρξει μια πλούσια διαδικασιών. Θα ήθελα κατά τα άλλα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί το έργο το οποίο πετέλεσε πραγματικά ήταν εξαίρετο και είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο γιατί με δυσκολία μπορούμε να καταλάβουμε εδώ περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάνν Μούλντερ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για τον ενθουσιασμό, το ζήλο που έδειξε για το ζήτημα αυτό. Έριξα μια ματιά στις τροπολογίες και η πρώτη εντύπωση που έχω είναι ότι το κείμενο, όπως προτείνεται, είναι πιο εκτενές πλέον. Δεν θεωρείται πλέον ότι ζητάμε πάρα πολλές λεπτομεριακές αλλαγές. Αν δω για παράδειγμα την τροπολογία 48, εδώ ζητείτε να υπάρχει ένας κατάλογος όλου του προσωπικού, όλων των αντιπροσωπιών εντός, εκτός των θεσμικών οργάνων. Ξέρετε ότι, για παράδειγμα, αν σε μια αποστολή στο Ναϊρόμπι υπάρχει ένας οδηγός ο οποίος προσλαμβάνεται ως εξωτερικό συνεργάτης, αυτό δεν με απασχολεί άμεσα, δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καταγράφεται με τέτοια αυστηρότητα. Όπως είπε άλλωστε και ο κύριος Σοντή... πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο ζήτημα της, του σφάλματος. Αποδεχόμαστε ούτως ή άλλως σε εθνικό επίπεδο ένα ποσοστό 2% όσον αφορά το σφάλμα. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό και πιστεύω θα πρέπει να διευθετηθεί σωστά είναι οι εθνικές δηλώσεις που γίνονται. Όταν ένα 80% των πόρων τυχαίων διαχείρισης από τα κράτη-μέλη τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλαμβάνεται και η σωστή πολιτική ευθύνη. Και νομίζω το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης θα πρέπει να διευθετείται και στα πλαίσια της διοργανική Συμφωνίας. Βλέπουμε ότι το Συμβούλιο στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής προσπαθεί να αποποιηθεί την ευθύνη αυτή. Και ένα ακόμα σημείο για το οποίο δεν είμαι απόλυτα σίγουρο. Πάντω, είχαμε πάντα ένα προπολογισμό ο οποίο πήγαινε από την 1η Ιανουαρίου ω τι 31 Δεκεμβρίου με μία μόνο εξαίρεση. Και αυτό ήταν για τη γεωργία, για τον γεωργικό τομέα, που η προθεσμία ήταν μέχρι τι 15 Οκτωβρίου και μετά τι 15 Οκτωβρίου ξεκινούσε το νέο οικονομικό έτο. Ισχύει ακόμα κάτι τέτοιο. Αν ισχύει όμω αυτό ακόμα, αν έχει παραμείνει, θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτά που ισχύουν στου υπόλοιπου τομεί. Ξέρετε ότι είχε προκύψει η κατάσταση αυτή γιατί υπήρχε μια στενότητα χρηματική τη δεκαετία του 80, δεν γίνεται όμως να συνεχιστεί η πρακτική αυτή. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πούμε κάτι ακόμα όσον αφορά τις πιστώσεις για τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Νομίζω ότι τα 200 δισεκατομμύρια τα οποία προτείνονται είναι υπερβολικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπονται πιο αυστηροί κανόνες έτσι ώστε να μην έχουμε πιστώσεις για να λείψει υποχρεώσεων οι οποίες δεν μπορούν να ισχύσουν, δεν μπορούν να αλλοποιηθούν γέρος. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πολύ Γιάν. Τώρα η Χέλγκα έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ Γιούτα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ίγκε για το έργο της και τις, την πληθώρα των προτάσεων της βελτίωσης. Και θα ήθελα να συγκεντρωθώ σε ένα σημείο, από την άποψή μου σημαντικό μέλος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, όσον αφορά το δημοσιονομικό, κανονισμό. Βρίσκω πολύ καλές προτάσεις της Σίγκε Γκρέσλε γιατί δικαιολογημένα επιχειρηματολογεί ότι πολλές φορές πρόκειται για ζήτημα αποδοχής. Ε, αυτό αφορά τον τομέα του πολιτισμού, για παράδειγμα μη κυβερνητικού οργανισμού που δεν έχουν πολλά κεφάλαια και πιέζουν εδώ και πολλά χρόνια όσο μικρότερα είναι τα ποσά τα οποία διατίθεται, τόσο μικρότερο είναι το διοικητικό άχθος. Το να λέγεται αυτό ε, ρητά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Και πραγματικά εύχομαι να διευκολύνουμε το έργο ε, των πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων γιατί εδώ και πολλά χρόνια πραγματικά ε, τις διώξαμε από κοντά μας γιατί τους εξενέβησε πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ τα θέματα αυτά που σχετίζονται με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι για το ανεκτό κίνδυνο, tolerable risk. Και νομίζω ότι η Ingeborg ε, έχει δίκιο, έχει δοκιμαστεί το μοντέλο αυτό διεθνώς και ε, θα ήταν καλό να έχουμε και κάποιες πληροφορίες από την, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν σχέση με τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες με αυτό το σύστημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό γιατί εάν γίνεται ο σωστός έλεγχος, η σωστή παρακολούθηση, ένα τέτοιο είδους εργαλείο που επιτρέπει ένα μικρό περιθώριο ελέγχου είναι ένα σωστό εργαλείο ενδεχομένω. Αλλά βεβαίω χρειαζόμαστε, όπω είπα, κάποιε επιπρόσθετε πληροφορίε εδώ. Ο Γιάννης Γκάιερ αναφέρθηκε στο θέμα του αρνητικού αποθεματικού ε, και με το διορθωτικό προπολογισμό τι θα πρέπει να γίνει εδώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας για να οριστικοποιήσουμε την άποψή μας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής έθεσε λίγο πολύ άμεσα κάποιες ερωτήσεις και νομίζω ότι θέλει μία απάντηση από την Ίγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω ξανά την κυρία Γκρέσλε για την παρουσίαση που μας έκανε και να την ευχαριστήσω και για την πολύ καλή συνεργασία, στενή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της όλης προετοιμασίας. Πέραν αυτού δεν συμφωνούμε βεβαίως για όλα και θα πρέπει εδώ να σταθώ σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Κάποιες γενικές λοιπόν παρατηρήσεις και μετά κάποιες ειδικότερε. Η γενική παρατηρήση είναι ότι ακούω πολλά στην Επιτροπή μας και στο Ευρωκοινοβούλιο γενικώ για μια γενική προτίμηση που υπάρχει για την απλούστευση. Συμμεριζόμαστε αυτόν το σκοπό. Όμως ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας ούτως ή άλλως οδεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις, κάποιες τροπολογίες οι οποίες δεν οδεύουν σε αυτή την οδό της απλούστευσης. να πω ας πούμε ότι παρόλο που σέβομαι απόλυτα τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου σε θέματα ελέγχου μου φαίνεται ωστόσο ότι η αποτελεσματικότητα θα προκύψει και εφόσον κάθε θεσμικό όργανο αναλάβει πραγματικά τις ευθύνες του και κρίνεται βάσει των όσων διενεργεί εντός κάποιου πλαισίου που είναι προκαθορισμένο και υπάρχει κάποιο περιθώριο διαχείρισης. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η Επιτροπή βρίσκεται σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα ανελαστικό. Ε, αυτό δεν είναι απλούστευση και το κόστος αυτό, αυτής της διαδικασίας επιβάλλει επιπλέον κόστη τα οποία δεν μπορεί μόνο να, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει. Εξελίσσονται όλε οι πολιτικέ μα ω προ τα διοικητικέ δαπάνε. και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξεχνούμε. Νομίζω λοιπόν ότι έχει προκύψει κάποια σύγχυση μεταξύ του στόχου από τη μια της απλούστευση και από την άλλη της ανάγκης να υπάρχει έλεγχος. Σημαντική ανάγκη δεν μπορώ να πω. Πρώτα απ' όλα για τα κάναμε μία πρόταση με στόχο να μειωθεί η γραφειοκρατία. Την πρόταση αυτή δεν την κάναμε στο κενό. Αυτό που προτείνουμε είναι να καθορίσουμε γραπτός το τι ακριβώς έχουμε κάνει μαζί από το 2009. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Όλοι νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο κατά τον οποίο υλοποιήσαμε τα μεταβατικά στοιχεία. Μεταβατικά στοιχεία για την ε, εκτέλεση και την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Γιατί να πάμε προς τα πίσω, γιατί να, να τρέξουμε στο παρελθόν. γιατί υπάρχουν διαδικασίε που λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Από την άλλη, ευχαριστώ την κυρία Γκρέσλι που αποδέχτηκε να φτάσει στο 15% το ποσό κάποιων μεταφορών. Μα ικανοποιεί αυτό παρόλο που δεν είναι αρκετό. Από την άλλη, θα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά το τέλο τη χρονιά, όπου δεν θα έχουμε καταφέρει κάποιε μεταφορέ να τι έχουμε περάσει κατεπηγόντω εντό των προθεσμιών που έχουμε ορίσει ή που έχουμε ορίσει εκ νέου. και η πρόταση τη εισηγήτρια εδώ κάνει τη διαδικασία αρκετά περίπλοκα και δεν μπορούμε να μεταμιεύσουμε κάποιε πιστώσει τη στιγμή που θα τι χρειαζόμαστε ή εγκαίρω. Σε ό,τι αφορά επίση τι επιδοτήσεις. Εδώ υπάρχουν κάποια όμορφα στοιχεία τα οποία τα δεχόμαστε με ευνοϊκά αλλά παραμένουν και κάποιες τροπολογίες που μας ανησυχούν. Εάν εγκριθούν θα αυξήσουν κατά τρόπο σημαντικό το φόρτο εργασία και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δικαιούχων σε μεγάλο βαθμό. Θα αντίκεινται στου στόχου απλούστευση. Να αναφερθώ εντάχει στο θέμα της Εσωτερικής Επιτροπής Clearing στον εξάμεινη προθεσμία για επιδότηση εντός της οποίας λύγει η διαδικασία ενός διαγωνισμού και την, ε, τα κριτήρια για την ανάληψη νομικών υποχρεώσεων. Η επιλεξιμότητα, η υποχρεωτική επιλεξιμότητα ε, για κάποια από τα κόστη και η τήρηση αρχείων. Μα είπε η κυρία Γκρέσλι ότι μπορούμε να περάσουμε στα 10 αντί για τα 5 χρόνια. 10 χρόνια είναι τεράστιο φόρτο για του δικαιούχου και για τα θεσμικά όργανα. Ο καθένας μας για τους λογαριασμούς ΔΕΗ τηλεφώνου ξέρει ότι τα κατάει το πολύ πέντε χρόνια. Πόσα αρχεία να βάλουμε στα ντουλάπια μας. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για διοικητικές αρχές, για δικαιούχους οι οποίοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτούς τους κανόνες. Σε μια δεκαετία Μερικοί από αυτούς ίσως και να έχουν ε, χαθεί. Πρόεδρε, δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση σε αυτή τη φάση. Απλώς να επισημάνω στα μέλη της Επιτροπής ότι υπάρχει το πρόβλημα της απλούστευσης. Και επειδή και ο κύριος Γιάγερ για τις μεταφορές ε, τράβηξε την προσοχή μου, να θυμίσω ότι υπάρχουν και κάποια στατιστικά στοιχεία για τους αριθμούς ε, που ζητήθηκαν και σχολιάστηκαν. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η Ίγκε για να ολοκληρώσει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά, αν τα πράγματα είχαν όπως λέτε, θα πρέπει να πάμε στα οδοφράγματα μαζικά και να μην εγκρίνουμε αυτή την έκθεση, καμιά της γραμμή. Ξέρω ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να κρατούν τα αρχεία τους 18 ή 20 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτό που οποίο προτείνουμε εδώ είναι μια ξεκάθαρη συντόμευση. Έχουμε δικαιούχους του κοινωνικού ταμείου που κρατάνε και για μικρότερα ποσά παραστατικά για 20 χρόνια, όπως σας είπα. Ε, δεν είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέτε, απλώς δεν αληθεύει. Και το ίδιο ισχύει και για ορισμένα τμήματα των μεταφορών. Και θα ήθελα πράγματι να σας επισημάνω ότι το ζήτημα της ε, απλούστευσης, πόση απλούστευση προτείνει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να το συζητήσουμε την ε, Παρασκευή σε μια προσεχή μας συνεδρίαση αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, λύνει απολύτως κανένα πρόβλημα με το Ταμείο. Λύνει το πρόβλημα της Επιτροπής μετακυλίοντας την ευθύνη από την Επιτροπή προς άλλους. Ε, και θεωρώ ότι δεν μου να το πράξει οι δικές μου τροπολογίες ε, προσπαθούν να διατηρήσουν ένα ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση των ευρωπαϊκών κοντιλίων. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ικανοποιητικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει απλώς, να περιοριστεί απλώς σε ένα δρό ρόλο εποπτείας ε, και στη συνέχεια να μας στέλνει το λογαριασμό ε, χωρίς ε, να αναλαμβάνει τελικά τις ευθύνες της. Ε, η δική μας πρόταση προσπαθεί να εφαρμόσει τη Λισαβόνα και μόνο τη Λισαβόνα. Προσπαθούμε να πετύχουμε κάποιες απλουστεύσεις, όπως για παράδειγμα τα έξι χρόνια τα οποία διαπιστώνουμε σε ορισμένα ταμεία ε, και βλέπουμε ότι ε, όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ ε, επικρατεί ένα κομφούζιο. Γι' αυτό θεωρώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια σαφήνεια. Γιατί συνήθως υπάρχουν και πάρα πολλές αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Εάν δεν ξεκαθαρίσουν όλα αυτά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω ε, και πάλι τονίσω τις προθέσεις αυτού του σχεδίου έκθεσης. Ε, προσπαθούμε τα νέα εργαλεία τα οποία έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσπαθούμε να τα αξιολογήσουμε και να θεσπίσουμε την ιδέα επίσης της δυνατότητας του ελέγχου, της ελεγξιμότητας αυτών των εργαλείων. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλουμε να περιοριστούμε στα υφιστάμενα εργαλεία. Αυτό το οποίο έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια με διάφορα εντελώς ετερογενή μεταξύ τους εργαλεία τα οποία εφαρμόζονται εντελώς ε, επιπόλαια και επιφανειακά ε, νομίζω ότι μια, ένας περαιτέρω πολλαπλασιασμός των εργαλείων αυτών και των μοντέλων ε, θα μας οδηγήσει σε ανυπέρβλητες δυσκολίες. Όσον αφορά τον ανεκτό κίνδυνο, ε, ε συζητήσαμε με την Επιτροπή, θεωρούμε ότι η Επιτροπή το έχει κάνει ένα εργαλείο για την απαλλαγή νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε, να συνεργαστούμε με την Επιτροπή εδώ ε, και με το ελεγκτικό ε, συνέδριο. Ε, γιατί έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία εδώ, γιατί δεν θέλουμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά θέλουμε να βασιστούμε στην υπάρχουσα εμπειρία μας η Σάντου λέει, ε, έχει δίκιο όταν λέει ότι έχουμε ένα τεράστιο χρονοδιάγραμμα για την απαλλαγή. Προσπαθήσαμε να το συντομεύσουμε, αλλά ό,τι και να κάνουμε, ε, ό,τι και να κάναμε δεν μπορούσαμε να παρακαιρδίσουμε ένα μήνα μόνο. Ε, δεν καταφέραμε τίποτα καλύτερο. εκτός αν κινηθούμε εντελώς ριζοσπαστικά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα κτίρια, θα ήθελα να συζητήσω με τη συνάδελφα κυρία Χολμάιερ. Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να κάνει κάποια χρέη μελλοντικά όσον αφορά την πολιτική των κτηρίων. Αυτό είναι το σκεπτικό εδώ. Ε, μελλοντικά δηλαδή δεν θα πρέπει να ε, προστρέχουμε στους ε, υφιστάμενους μηχανισμούς χρηματοδότησης, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια χρέη. Εδώ θα γίνει σκληρή διαπραγμάτευση. Τώρα, αγαπητέ Γιάννη, νομίζω ότι οδεύουμε προς ένα συμβιβασμό. Ε, την Παρασκευή θα έχουμε ένα γύρο συζητήσεων με την Επιτροπή. Θα επιστρέψουμε ενισχυμένοι από το Παλέρμο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι εδώ. τώρα, για τον συνάδελφο κ. Μούλτερ, αυτές οι τροπολογίες για το άρθρο 48, δεν πρόκειται για μια τροπολογία εδώ, αλλά αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και το τι διαπραγματευθήκαμε με το Συμβούλιο. Και θεωρώ θα πρέπει να παραμείνει. Πρόκειται για μια παλιά ιστορία η οποία εδράζεται σε μια πλατιά συνένεση. πέτυχε και ο συνάδελφο κ. Γκαλτιέρη Εγώ ίδια έχω παρουσιάσει κάποιες ε, άλλες ε, τροπολογίες όσον αφορά το προσωπικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία εποπτεία. 45.000 ε, μόνιμους υπαλλήλους, αλλά στο, στα ταμεία της Κομισιόν υπάρχουν ε, είναι εγγεγραμμένα 66.000 άτομα. Ε, δεν ξέρουμε πώς είναι τα... ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ε, απασχολούμενων, των εργαζόμενων εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, από την απαλλαγή περιμένουμε μια πλατιά αλλαγή αλλά οι αλλαγές αυτές δεν έχουν για το τρέ... σημασία για το τρέχον έτος. Τώρα, για την κυρία Τρούπελ, όσον αφορά την διαγραφή του αρνητικού αποθεματικού, υπάρχει μια σχετική τροπολογία και τον περιορισμό επίσης των διορθωτικών επιστολών. Ε, υπάρχει εδώ η σχετική τροπολογία. Ε, νομίζω πρέπει να περιοριστούμε εδώ σε μία ή δύο διορθωτικές επιστολές, να μην επεκταθούμε σε περισσότερες. Θεωρώ ότι θα είναι καλό για την πειθαρχία μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω την ε, Παρασκευή να επιτευχθούν κάποιοι συμβιβασμοί εκεί που κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Αλλά ε, νομίζω ότι για το Παλέρμο δεν έχεις δίκιο. Τώρα, χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο για αυτό το σημείο της της διάταξης, πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι υπέθεσα. Και τώρα έχουν φτάσει εντωμεταξύ όλοι μας οι προσκεκλημένοι για το σημείο της της διάταξης που αφορά την μελέτη. Και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή και ο εισηγητής ήδη δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να μετακινήσουμε τα, το, τα σημεία του Ράιμερ μετά την παρουσίαση του Ράιμερ Μπέγκε, το πακέτο Μπέγκε να ακολουθεί στην παρουσίαση της μελέτης. Και τώρα καταρχήν να ακούσουμε, να συζητήσουμε μάλλον τη μελέτη. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να συζητήσουμε αυτή τη ε, μελέτη που μας απασχόλησε εξάλλου. Νομίζω ότι αυτό είναι συνηθισμένο εδώ. Ε, ε, προκρίθηκε με το συνηθισμένο τρόπο και κάποιος εξωτερικός ε, επιστήμων ανέλαβε, κέρδισε αυτό το διαγωνισμό και ανέλαβε αυτή τη μελέτη αλλά στη συνέχεια υπήρξαν κάποια σημεία τριβής. Γι' αυτό θα εφαρμόσουμε την εξής διαδικασία οι δύο συνάδελφοι, στην περίπτωση αυτή δύο άνδρες συνάδελφοι, οι δύο αντιπρόεδροι που ήταν αρμόδιοι για αυτή την επιτροπή θα κάνουν μια σύντομη παρουσίαση γιατί και εδώ προβλέπεται μόνο μια ώρα. Θα μας κάνουν μια σύντομη εισαγωγή, μια σύντομη παρουσίαση αυτής της ε, μελέτης και στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο του Λίτς τη μελέτη και τα αποτελέσματά της και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο αυτοί που επιθυμούν να το πράξουν. Ο, προ... ο Φίλιπ Μάινστατ, ο εκπρόσωπος της EBRD, ο Γιάνν Φίσερ και ο κύριος ε, Τόμας θα πάρουν το λόγο και στη συνέχεια θα περάσουμε στην ε, γενικότερη συζήτηση και ο Ιάλο κάλφιν είναι ο Ιβάλο, κάποιος, ο Ιβάλο Κάλφιν σε αυτή την περίπτωση, ο οποίος θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ο Ιβάλο Κάλφιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η βασική ιδέα όταν ζητήσαμε να γίνει η μελέτη αυτή ήταν ε, να μπορούμε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα τα οποία είχαν ανακύψει κατά τη διάρκεια συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν είδαμε ότι υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ζητήματα όπως η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, η πολιτική για την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδυτικά προγράμματα όπως το ΙΤΕΡ και τον Καλλιλέο, από τη μια λοιπόν πολιτική βούληση για τα αισθήματα αυτά και από την άλλη περιορισμένη δημοσιονομική πόρη στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι πολιτικοί αυτοί στόχοι τους οποίους συζητούσαμε. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, Είδαμε ότι ε, εκτελήθηκε και μία εθνική συζήτηση όσον αφορά τα μέτρα λιτότητα, τα οποία έχουν ληφθεί πλέον σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στι συζητήσει του κοινοτικού προπολογισμού, αλλά και σε όλε τι συζητήσει που γίνονται για τι εθνικέ αναλήψει ε, υποχρεώσεων όσον αφορά την ε, επίτευξη των κοινοτικών στόχων από τα κράτη-μέλη. Το ζήτημα το οποίο συζητήσαμε στο παρελθόν και το συζητάμε και σήμερα είναι ακριβώς αυτό, η έλλειψη δημοσιονομικών πόρων για την επίτευξη των πολιτικών στόχων, ζήτημα το οποίο συνδέεται και με την δυνατότητα αύξησης των ιδίων πόρων του κοινοτικού προπολογισμού, καθώς επίσης και την ε, δυνατότητα να έχουμε τη δυνατότητα προσέλκυσης επιπλέον πόρων και επένδυσης των πόρων αυτών. Οι δυνατότητες όσον αφορά τη δυνατότητα μόχλευσης μπορεί να έρθει μόνο μέσω της ε, συγχρηματοδότησης, κοινοτική δηλαδή και εθνική πόρη, αλλά και μέσω της δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Ακούστε και όμως και δυνατότητα να συνεργαστούμε περισσότερο με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδίω με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι άλλωστε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια τράπεζα αυτή καθ' αυτή για τι επενδύσει οι οποίε γίνονται στα κοινοτικά προγράμματα. Είπαμε ότι θα έπρεπε να συνεργαστούμε όμω και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Στόχο μα λοιπόν ήταν να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση αυτή για να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουμε για να αυξήσουμε την συμμετοχή όλων των υπόλοιπων μέσων τη ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων. Οι επιπλέον αυτοί πόροι θα μπορούσαν να έρθουν από πολλέ και διάφορε πηγέ και σίγουρα η ακολουθητή διαδικασία θα είναι πολύπλοκη. Ωστόσο, γίνονται ήδη κάποιε προτάσει από τι ίδιε τι τράπεζε. Πρόσφατα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είδαμε μια παρουσίαση του κύριου Μέιστατ για το, τα λεγόμενα European Project Bonds, ευρωπαϊκά ομόλογα για συγκεκριμένα κοινοτικά έργα, που είπαμε ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν εν μέρη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήσαμε και σε άλλες επιτροπές το ζήτημα αυτό και σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε μια επίσημη απόφαση. Για την έκθεση ακολουθήθηκε μια πολύ διαφανής διαδικασία. Απευθυνθήκαμε σε εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τα πορίσματα της μελέτης. Η μελέτη αυτή βέβαια περιλαμβάνει τη δική τους άποψη όσον αφορά το ζήτημα αυτό το οποίο αποτέλεσε το αντικείμενο της μελέτης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μελέτη αυτή ως μία απλώς πηγή α, περαιτέρω ιδεών, πληροφόρησης που θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφου, συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμμετείχανε στην θέσπιση του πλαισίου για την εκπόνηση της μελέτης αυτής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες βέβαια της μελέτης και θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που είναι πάντα παρόντες στις συζητήσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθούν μαζί με εμά να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τίθενται. Θα, δεν θα ήθελα να αναλώσω περισσότερο χρόνο, κυρία Πρόεδρε. Εδώ έθεσα το γενικότερο πλαίσιο της μελέτης αυτής και θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στους ίδιους συντάκτες της μελέτης και θα έχουμε δυνατότητα βέβαια να υποβάλουμε και ερωτήματα και παρατηρήσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ρόμπινσον και τον κύριο Πέιτ να μας παρουσιάσουν την μελέτη. με ακούτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε και μου αρέσει πάρα πολύ κιόλα ε, να στέκομαι για να μιλήσω σαν καθηγητής. Δυσκολεύομαι να παρουσιάζω καθιστώ. Αυτό που θα κάνω λοιπόν σήμερα είναι να διατρέξω ε, με, εν συντομία τα πορίσματα της μελέτης για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και με τα μέλη της Επιτροπής σας. Εγώ και ο συνάδελφος θα παρουσιάσουμε από κοινού τα πορίσματα της μελέτης και πολύ γρήγορα θα σας ε, συστηθούμε και θα επικεντρωθούμε στις συστάσεις και τα συμπεράσματα. Όμως θα δούμε θέματα του πλαισίου, να σας εξηγήσουμε τι εννοούμε με τη συγχρηματοδότηση και κάποια βασικά ζητήματα. Θα σας πω πώς, τι μεθοδολογία ακολουθήσαμε για τα πορίσματά μας και θα παραμείνω όπως προείπα στα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Now, Σύντομα, να σας πω ότι εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Είμαι καθηγητής οικονομικών και δημόσιας πολιτικής εδώ και 10 χρόνια. Έχω κάνει πολλές δημοσιεύσεις και συμβουλευτικό όργο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ενδιαφέρει ιδιαίτερω η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από τον ακαδημαϊκό κόσμο αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερω μάλιστα πολιτική δαπανών. Κάτι που σας ενδιαφέρει και εσάς εδώ ιδιαίτερως, αλλά και στην ε, ακαδημαϊκή μας πρακτική. Να δώσω το λόγο και στον συνάδελφο για να παρουσιαστεί. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Το όνομά μου είναι Ρόμπερτ Μπέιν. Είμαι ανεξάρτητος ε, σύμβουλος για θέματα οικονομικών και ως προς τη συγκεκριμένη μελέτη και εγώ έχω συνεργαστεί συμβουλευτικός και με την Τράπεζα Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαι βοηθό καθηγητή, μάλλον είμαι researcher fellow, δηλαδή ερευνητή ανεξάρτητος στο Πανεπιστήμιο του Λίτ και έχω εργαστεί ως σύμβουλο εταιρείε μεταφορών και συγκοινωνιών. Πολύ γρήγορα το πλαίσιο τη μελέτης πριν περάσω στα ερευνητικά ζητήματα που μας απασχόλησαν. Πρώτα απ' όλα, να ορίσουμε τι εννοούμε με τη συγχρηματοδότηση για το πλαίσιο της έρευνάς μας. Μιλάμε για δανειοδότηση εκτός δωρεών. Μιλάμε για χρήματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από την Τράπεζα Ανάπτυξης. Εδώ η συγχρηματοδότηση που μας ενδιαφέρει είναι ακριβώς αυτή, αλλά το ποσοστό είναι πολύ μικρό. 1% του συνολικού προπολογισμού που αποδίδεται κατά αυτόν τον τρόπο σε δικαιούχους. Θα δούμε πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον με τα απορίσματα της έρευνά μας. Και Σύμφωνα και με άλλε πολλέ μελέτε που έχουν εξετάσει τη χρηματοδότηση και την, ε, το συνδυασμό πολλών διαφορετικών μεθόδων, βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστιο περιθώριο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανατρέξει περισσότερο από το όργανο χρηματοδότηση στο μέλλον. Υπάρχει τρόπος με οικονομικούς διαμεσολαβητές να συνεργαστούμε ώστε και με άλλους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς να πάρουμε ένα μέρος από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και να, μετακινήσουμε από εκεί το φόρτο, το άχθος. Ε, επίσης μπορεί να έχουμε εμπορικούς δανειστές της αγοράς μάλιστα και έτσι και αυτοί να αναπτύξουν ευρωπαϊκούς στόχους και ευρωπαϊκές προτεραιότητες μέσω αυτών των εργαλείων. Um, Πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω το πρώτο σύνολο των ερευνητικών ζητημάτων που, μας ζητήθη, που καλέσαμε τους αυτούς μας να απαντήσουμε. Πρώτα απ' όλα για, την, ε, για το δημοσιονομική λογοδοσία. Αναρωτηθήκαμε κατά πόσον οι δύο τράπεζες, η EIB και η ERD, ε, μπορεί να αναλάβουν ευθύνε σε περίπτωση που υπάρχουν αποτυχίε στι δανειοδοτικέ διαδικασίε. Και έπειτα ασχοληθήκαμε με την εξωτερική εντολή τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τον συγκεκριμένο μηχανισμό ε, ταμείευση ε, που κάποιοι γνωρίζουν, τουλάχιστον στου γενικού του όρου. Και επίση το τι κανόνε και τι προστασία μπορεί να συνδυαστούν για τον ώστε να ωφεληθεί ο ευρωπαϊκό προπολογισμό του σημερινού του σχεδιασμού. Κατά τρίτον, και ως προς τις εγγυήσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, να ζητήσαμε τι δυνατότητες δημοσιονομικής διαχείρισης υπάρχουν, ώστε να έχουμε εκτεταμένη χρήση της χρηματοδότηση ενδεχομένως, προκειμένου να πετύχουμε μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία. Εδώ θα γίνει μια διάκριση μεταξύ της άμεσης χρηματοδότησης, ε, μάλλον άμεσης δανειοδότησης μάλλον προς τα κράτη-μέλη και τη έμεση. με ευρωπαϊκές εγγυήσεις ή και με τι δανειοδοτήσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προ τρίτε χώρε. Επίσης, να σας πω ότι είδαμε και κάτι που ίσως έχει και περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα, μια σειρά ζητημάτων. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι η όρια αναφορά εδώ ήταν πολύ καθοριστική σημασία, γιατί ε, ε, έγιναν πολλά, έγιναν πολλά ερωτήματα. Και μας απασχόλησε και η κοινοβουλευτική αναθεώρηση κάποιων από τις διαδικασίες που μελετήσαμε εδώ, όπως έχουν εξελιχθεί ως τώρα. Τώρα, από την αρχή αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι να διακρίνουμε μεταξύ επίσημων μηχανισμών και θεσμικών διαδικασιών που υπάρχουν για τον έλεγχο σε αντίθεση με άτυπες πρακτικές και πώ ακριβώ λειτουργούν ε, αυτέ οι διαδικασίε, Δηλαδή από τη μια έχουμε το τι λέει η συνθήκη και το τι συμβαίνει στην πράξη. Πολλέ φορέ δεν ήταν απλό να διακρινώ μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών φαινομένων. Ε, εξαιρετική σημασία στο σημερινό πλαίσιο είναι ο βαθμό κατά τον οποίο τα όργανα αυτά θα μα επέτρεπαν να πετύχουμε, να επιδιώκουμε του ευρωπαϊκά στρατηγικούς στόχου. Και υπάρχει και μια σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν ως προ τη συνεργασία με την τράπεζα Ιδίω επειδή χρειάζεται δανειστή για να παράσει τα κονδύλια και θέτει κάποιους όρου για τα αποτελέσματα που επιδιώκονται. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μα απασχολήσει. Η διακυβέρνηση και η διαφάνεια, αυτά είναι πολύ διαφορετικά για μας από ότι η προβολή, διαχείριση εδώ, η διακυβέρνηση αναφέρεται στο βαθμό που οι διαθεσμικέ σχέσει επιτρέπουν ε, πρόσβαση στο κοινό εάν υπάρχουν ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες που μπορεί να ενδιαφέρουν και το Ευρωκοινοβούλιο ως προς τον τρόπο που εξελίσσονται, αλλά και μεταξύ τραπεζών μεταξύ τους, ε, μεταξύ των τραπεζών των ιδίων μάλλον, όπου μπορεί να υπάρχουν ε, θέματα εμπιστευτικότητας, θέματα διαφάνειας. Όλα αυτά διαφέρουν από την προβολή, από καθώς όλοι θα γνωρίζετε αυτό το πρόβλημα είναι διαρκές στις οικονομικέ δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που χρειάστηκε όμω να κάνουμε εμείς είναι να ξεχωρίσουμε τις επιπτώσεις της χρηματοδότηση για την προβολή ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μεταξύ των πολιτών και των δικαιούχων, αλλά και το τι συμβαίνει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κάτι που κάνει και τη δουλειά του Κοινοβουλίου πολλέ φορέ πιο δύσκολη. Ω προ την κατανόηση του τρόπου κατά τον οποίο διοργανώνεται ο ίδιο ο ε, προπολογισμό. Κάποιε φορέ πώ ε, κατακαιρματίζεται και πώ τελικά δαπανάται. Εδώ λοιπόν συνδυάσαμε τρει κλασικέ μεθόδου. Πρώτα απ' όλα μελετήσαμε όλε τι υπάρχουσε μελέτε σε αυτόν τον τομέα, τι συγκεντρώσαμε γιατί έχουμε και οι δυο μα ερευνητέ 30 ετή πήρα πίσω μα και συνομιλήσαμε τουλάχιστον με 50 άτομα και από τις δύο τράπεζες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Ήταν πολύ χρήσιμες συζητήσεις αυτής, ε, αυτές για μας και ήταν ε, πολύτιμη η στήριξή τους. Βέβαια πήραμε πολλές αντιφατικές απαντήσεις και είχαμε και αντιφατικά συμπεράσματα. Οπότε όταν θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε το κείμενο θα το καταλάβετε. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι είναι στα πορίσματα αυτά να προσφέρουμε και τη δική μας ακαδημαϊκή γνώση ώστε να γίνουν αξιοποιήσιμα τα πορίσματα αυτά. Ως προς τη διάρθρωση της ε, έκθεσης, όπως θα φαντάζεστε, υπάρχει ένα κεφάλαιο μετά την εισαγωγή που εξηγούμε τι κάνουμε για τις δύο τράπεζες τις ίδιες, με μια περιγραφή, ποιες είναι οι διαφορές τους, ποιες οι ομοιότητες εκτεταμένα γίνεται λόγο για τη σωματοδότηση εντό Ευρωπαϊκή Ένωσης. Στο κεφάλαιο 4 ασχολούμαστε με τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, το θέμα της εξωτερικής εντολής, το θέμα των ε, δανειοδοτικών εγγυήσεων προς τα κράτη-μέλη και μετά συμπεράσματα και συστάσεις. Είναι εκτεταμένο και το παράρτημα ουσιαστικά ελέγχει, εξ, αποτιμά όλα τα υπάρχοντα εργαλεία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο τμήμα του εγγράφου συνολικά. Ελπίζω ότι θα αποδειχτεί να είναι και στην πράξη χρήσιμο. Θα ήθελα να καταφέρω στα επόμενα 5 10 λεπτά να συνοψίσω λίγο την όλη μελέτη. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα σημαντικότερα σημεία. Το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι ο κοινοτικό προπολογισμό όσον αφορά τη χρηματοδότηση δεν δημιουργεί κανένα άμεσο κίνδυνο όσον αφορά το μέγεθος της χρηματοδότηση και τον τρόπο διεξαγωγής της. Βλέπουμε ότι γίνονται συγκεκριμένε διαθεσιμότητες πιστώσεων σε συγκεκριμένα έργα και δεν υπάρχει καμία πλέον εγγύηση πέρα από τη συγκεκριμένη αυτή δέσμευση. Όσον αφορά τώρα την εξωτερική εντολή και το ζήτημα του Ταμείου Εγγυήσεων για την Εξωτερική Δράση, καταλήγουμε πολύ θετικά και εδώ πέρα ότι ευθυγραμμιζόμαστε εδώ πέρα ουσιαστικά με βορίσματα άλλων μελετών και ξέρετε ότι υπήρξε και μία πλήρης μελέτη όσον αφορά το Ταμείο Εγγυήσεων που είχε γίνει το 2010. και στα πλαίσια της μελέτης αυτής γίνανε πολλές ποσοτικές αναλύσεις και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα πρότυπα αναλύσεων του κινδύνου. Και το 2010 το ελεγκτικό συνέδριο και αυτό τοποθετήθηκε πολύ θετικά για τον τρόπο διαχείρισης του Ταμείου Εγγύσεων. Με λίγα λόγια λοιπόν, πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα πολύ κατάλληλο μέσο το οποίο προστατεύει τον προπολογισμό και τροφοδοτείται με πιστώσεις πολύ σωστά και καταλήλως μέσω του target rate του αστόχου του 9%. Να σας δείξω γρήγορα και μια διαφάνεια. Με κίτρινο βλέπετε την εγγυημένη δανειοδότηση, τη δανειοδότηση η οποία καλύπτεται από το Ταμείο Εγγυήσεων. Στα αριστερά το βλέπετε αυτό με τις κάθετες στήλες. Για παράδειγμα το 2009, τέλος του 2009, μιλάμε για 16 δισεκατομμύρια ευρώ δανειοδότηση το οποίο καλύπτεται από το Ταμείο Εγγυήσεων στα δεξιά, στην κάθε τη στήλη, βλέπετε τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το ταμείο αυτό και υπάρχει εδώ πέρα ένα μικρό σφάλμα στη διαφάνεια. Θα έπρεπε στα δεξιά να λέγεται billion, δισεκατομμύρια και όχι εκατομμύρια, γιατί μιλάμε εδώ για 1,3 δισεκατομμύρια για τα τέλη του 2009. Συνδυάσουμε τα δύο αυτά αριθμητικά στοιχεία, καταλήγουμε σε ένα ποσοστό 9% όσον αφορά την απόδοση από τις επενδύσεις αυτές και στις αρχές του 2011 έχουμε 140 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν και αυτά στο ποσοστό διάθεσης 9%. Περνάμε τώρα από το Ταμείο Εγγύσεων στις εγγύησεις προς τα κράτη-μέλη. Έχετε εδώ πέρα ένα μέσο το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντί να προβλέπονται συγκεκριμένε πιστώσεις για το μέσο αυτό, προβλέπεται στον προπολογισμό αυτό το οποίο ονομάζουμε περιθώριο, margin. Και θα ήθελα να δείξω στα μέλη εδώ πέρα της Επιτροπής ότι υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο ακόμα και για τον τρέχοντα προπολογισμό. Πρόκειται λοιπόν για ένα μέσο το οποίο δεν απειλεί σε καμία περίπτωση τον κοινοτικό προπολογισμό, δεν θέτει κανένα πρόβλημα, κανένα κίνδυνο και ούτε δημιουργεί εμπόδια στον τρόπο λειτουργία του Ταμείου Εγγυήσεων. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μέσο αυτό. Να σας ένα παράδειγμα. Έχω πάρει το 2011. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πλαφόν για τους ιδίους πόρους, 23% του ΑΕΠ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 152 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό το οποίο προβλέπεται για το φετινό έτος είναι 126,5 δισεκατομμύρια, 1,09% του ΑΕΠ του ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πέρα δημιουργείται ένα περιθώριο της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ και το περιθώριο αυτό καλύπτει πάρα πολλές περιπτώσεις εγγυήσεων όσον αφορά περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Έχετε εδώ πέρα επικαιροποιημένα στοιχεία από τους εξωματούχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι περνάνε στο σύστημα αυτό, στον πίνακα αυτό, όλα τα νέα ποσά που φτάνουν κάθε χρόνο. Μπορεί να έχουν τροποποιηθεί ενδεχομένω τα ποσά από τότε που συντάχθηκε ο πίνακα αυτό το Φεβρουάριο, οι αρχέ όμω παραμένουν οι ίδιε. Έχουμε εδώ πέρα τι πληρωμέ, αυτέ καθ' αυτέ έχουμε τι πληρωμέ που γίνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου στα χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έχουμε τι πληρωμέ που γίνονται μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δανειοδοτήσεων και έχουμε έπειτα και τη δανειοδότηση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προ τι τρίτε χώρε και το διαθέσιμο ποσό το οποίο έχετε είναι 25 δισεκατομμύρια ευρώ, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο για επιπλέον ποσά, το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και μεγαλύτερης ανταπόκρισης, αν θέλετε, σε κάποιες έκτες περιπτώσεις που προκύπτουν. Uh, Οι τελικές παρατηρήσεις αφορούν περισσότερο το πολιτικό σκέλος της όλης εξίσωσης, για να το πω έτσι. Το τελικό μέρος λοιπόν της μελέτης επαναλαμβάνει κάτι που ε, το ανέφερε προηγουμένω και ο Ρόμπι. Είναι 200 σελίδε η έκταση της, του ολοκειμένου. Δεν μπορώ να σα πω όλε τι λεπτομέρειε προφανώ, αλλά για τον έλεγχο του προπολογισμού. Είδαμε να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί έλεγχου και επίσημοι μηχανισμοί που δημιουργούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η όλη διαδικασία αυτή εμπλέκει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως ζητήματα που προκύπτουν και ανεπισήμως. Αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό και θετικό από τη θετική άποψη. Το γεγονός ότι τα ίδια τα δάνεια πρέπει να επιστραφούν, αυτό δημιουργεί μηχανισμούς ε, πειθαρχίας από της ουσίας υπάρχουν συστήματα τα οποία βασίζονται στην εκτέλεση εντολών και την πειθαρχία με τα όρια που δίνονται και των παραγγελιών επίσης, όμως υπάρχουν και πολλοί οικονομικοί διάμεσοι, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν και αυτά τα δικά τους τα συμφέροντα και να επηρεάζουν τον ε, έλεγχο των ε, ευρωπαϊκών φορέων. Η ευελιξία επίση είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλά από αυτά τα εργαλεία ε, που έχουν πολλές διαφορετικές μορφές και το κατά πόσο αυτά τα ίδια είναι ελαστικά μπορεί να κάνει την κατάσταση πιο απλή ή πιο περίπλοκη. Το συμπέρασμα που σας δίνω εδώ είναι κάπως ατελές, όμως υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη για διεξοδικότερη μελέτη για το τι ακριβώ συμβαίνει στην πράξη. έχει γίνει έρευνα για ένα από τα δυο αυτά εργαλεία θεωρητικά, αλλά δεν υπάρχει διεξοδική έρευνα που γίνεται στην πράξη. Αυτό είναι μια ανάγκη που ενδιαφέρει νομίζω τα μέλη της Επιτροπής σας. Τώρα, για τη συγχρηματοδότηση, πολλά είναι τα ωφέλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την άποψή μας και πιστεύουμε ότι ως μέθοδος αυτή είναι συμβατή με τους ευρωπαϊκούς στόχους γενικότερα. Δύο από τα εργαλεία που διεξοδικότερα ελέγξαμε μας οδήγησαν σε επαλήθευση των ε, συμπερασμάτων ε, και για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης Είδαμε την εταιρική σχέση για την επιχειρηματικότητα με πολύ καλά αποτελέσματα και είδαμε να υπάρχει και μια ισχυρή επιθυμία από τις ίδιες τις τράπεζες να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Οι τομείς που μας απασχόλησαν, που και εσείς θα πρέπει να εξετάσετε πολύ σοβαρά, είναι εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες επικαλύψεις μεταξύ των διαφορών εργαλείων Μάλιστα, επανειλημμένες επικαλύψεις μεταξύ των, ε, του, Τζέρεμι και των προγραμμάτων ΣΥΠ. Ε, αυτό το έχουν δει και άλλες μελέτες εκτός από τη δική μας. Ένα άλλο ζήτημα που είναι αρκετά προβληματικό είναι το κατά πόσο τα εργαλεία αυτά στα νέα κράτη-μέλη δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όπως το RSFF ή το ΣΥΠ. Δεν ξέρουμε κατά πόσον δίνει αποτελέσματα στα νέα κράτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το άλλο ζήτημα για του στατικικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά πόσον υπάρχει συνεργασία με τι διαφορετικέ τράπεζε και τι δυσκολίε μπορούν να προκύπτουν εδώ. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να διερευνήσουμε κάποιε μάλλον δεν έχει διαφορά το αν συνεργάζεται κανεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή κάποια άλλη από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Δεν είναι τόσο τεράστιες οι διαφορές μεταξύ των δύο τραπεζών. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του όλου έργου που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτελεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει επίσης τέτοια διάθεση γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρά ωφέλη. Το πώ λοιπόν μπορεί να υπάρξει καλύτερη συνεργασία με αυτέ τι δύο τράπεζε νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για εσά. Τα λέω όλα αυτά με πολύ περισσότερε λεπτομέρειε στο κείμενο. Για τα πολιτικά αποτελέσματα τώρα. Συνδυάσαμε εδώ κάποιε μελέτε περιπτώσεων, case studies, με τη γενική θεωρητικότερη συζήτηση και καταλήξαμε πάλι σε κάπως ανάμεικτα πορίσματα, αν μπορώ να τα πω έτσι. Υπάρχουν κάποια πραγματικά εντυπωσιακά θετικά αποτελέσματα ως προς τις προτεραιότητες της διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια λόγου χάρη, όπως την ανάγκη μεγαλύτερη συμμετοχή των 100 μέσω των προγραμμάτων Jasper. Αλλά σταθήκαμε και σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα πόσο αντίκτυπο λόγου χάρη έχει η οικονομική κρίση για τα νεα κατημέλη. Τα Jaspers έχουν δώσει καλά αποτελέσματα, όπω είπαμε, σε ορισμένα προγράμματα εκεί, αλλά παραμένουν μέγιστα προβλήματα απορρόφηση των κονδυλίων στα νεα κατημέλη. Το ερώτημα λοιπόν που παραμένει είναι το κατά πόσο η οικονομική κρίση μπορεί να έβλαψε την ε, αποδοτικότητα των ε, δημοσιονομικών εργαλείων. Αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Και υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, γι' αυτό θα επανέλθω στο ζήτημα του κατά πόσο έχουν αρκετά ανεπτυγμένε αγορέ τα νεα κράτη-μέλη ώστε να ανταποκριθούν στι ανάγκε τη χρηματοδότηση. Αυτό ανέκυψε πολλέ φορέ ε, στα συμπεράσματά μα. Τέλο, η διαφάνεια αρχικά πιστεύουμε ότι είναι περίπλοκο ζήτημα ώστε να το αντιμετωπίσει κανείς ολοκληρωμένα. Οι τράπεζες καταλαβαίνουν την ανάγκη της εμπορικής ε, εμπιστευτικότητας, όμως και το Ευρωκοινοβούλιο έχει τεράστια ανάγκη να έχει ε, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα το πώς, το, πώς εκταμιεύονται τα κονδύλια και πώς πανώνται. Εδώ λοιπόν όλα αυτά εμπλέκονται με το όλο θέμα της ε, διαφάνειας το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ετοίμασε δύο εκθέσεις φέτος, ε, τουλάχιστον για το θέμα της διαφάνειας και για το πόσο η διαφάνεια μπορεί να αφορά και τη χρηματοδότηση. Εδώ πρέπει να έχουμε και κριτικό πνεύμα δεν εννοώ να είναι κανείς επικριτικός προφανώς, εννοώ να έχει κριτική σκέψη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται σε ένα βαθμό να μην το έχει πράξει αυτό. Μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα με την αιμονή που έχει στη κρίση συγκεκριμένων εργαλείων, αλλά λίγη κριτική σκέψη δεν θα βλάψει. Και τέλος η προβολή. Είπα ότι αυτό είναι ένα διαρκέ πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει προκαλέσει πολλή σύγχυση ω τώρα και απογοητεύσει διότι δεν υπάρχει αρκετή προβολή των ευρωπαϊκών δαπανών και σίγουρα αυτό είναι απογοητευτικό. Αλλά μπορεί να προκύψουν και άλλοι προβληματισμοί και δυσκολίες ακόμη οξύτερες στο μέλλον, διότι τα ίδια τα εργαλεία όταν κανεί εργάζεται και συνεργάζεται με οικονομικού διαμέσους, ίσω να μην είναι τόσο σαφή για τον δικαιούχο πλέον, ακόμη περισσότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα διαφορά βαθμού μόνον, αλλά διαφορά είδου. Δηλαδή για τις ευρωπαϊκές δαπάνες δεν είναι μόνο στη συγχρηματοδότηση φανερό ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά συμβαίνει και σε όλα τα άλλα τα σκέλη της, του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ε, και για τα προγράμματα ΣΥ που σας υποτιμελετήσαμε κάτι τέτοιο ίσχυε. Επίσης, Σαφώ υπάρχουν επικοινωνιακέ δυσκολίε και δικέ μα προτάσει δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να υλοποιηθούν, αλλά ένα πρώτο πρακτικό βήμα θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια να γίνει πιο τολμηρή, να, να λάβει πιο καινοτόμε λύσει στα θεσμικά τη προβλήματα. Και όσοι συζήτησαν μαζί μα, παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν κάποιε δυσκολίε στη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, ας πούμε στη διαδικασία της χρηματοδότησης. Πολλά, πολλές δυσκολίες παραμένουν σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Τα συνολικά μας συμπεράσματα ήταν ότι το θέμα αυτό είναι συναρπαστικό. Πολύ τη ευχαριστηθήκαμε τη μελέτη στην διεξαγωγή τη. Ήταν μια πραγματική πρόκληση για μα ερευνητική. Όμω θα σα έλεγα εδώ να κάνουμε ένα αντάλλαγμα. Να, να προσπαθήσουμε δηλαδή να <clears throat> σκεφτούμε το τι γίνεται με τους απλοποιημένους δημοσιονομικούς μηχανισμούς σε σχέση με τον έλεγχο τις πολιτικές δυσκολίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσω πίσω τη σκητάλη στα δικά σας έμπειρα χέρια και θα σας αφήσω εσείς να δώσετε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα που παραμένουν μετά την παρουσίαση της μελέτης. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι για όλους όσους συνόδευσαν ευθύ εξ αρχής αυτή τη μελέτη, τα όσα ακούσαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και νομίζω ότι εδώ σε αυτή την Επιτροπή όταν ζητάτε ορατότητα, διαφάνεια και έλεγχο νομίζω ότι βρίσκεται πλατιά αποδοχή. Όσον αφορά την ορατότητα, την προβολή προσπαθούμε να την αυξήσουμε αλλά καμιά φορά προσκούμε πάνω σε γρανίτη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί μαζί μας όταν το ζητούμενο είναι να θεσπιστούν κάποια μέτρα τα οποία αυξάνουν την ορατότητα. Ε, ε, και μια, ε, νομίζω ότι εδώ μια ενιαία στρατηγική επικοινωνία θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Τώρα όμως έχουν το λόγο οι προσκεκλημένοι μας πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Ο πρόεδρος κύριος Μάλστο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω την μελέτη που μόλις μας παρουσιάστηκε. Θα έλεγα ότι δεν μπορώ να δεχτώ το να επιβεβαιώνουμε ότι ε, όλα αυτά τα σχόλια τα οποία γίνονται δεν ε, είναι βάσιμα. Εμείς, εφόσον μας το επιτρέπετε, μπορούμε να συμμετέχουμε σε μία συζήτηση η οποία θα σας δώσει και συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς επίσης και συγκεκριμένα δεδομένα προκειμένου να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας. Ωστόσο θα ήθελα να επικεντρωθώ στο βασικό ζήτημα το οποίο είναι το ακόλουθο. Να δούμε τελικά αν συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει το συνδυασμό πόρων από τον κοινοτικό προπολογισμό και πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κατά την άποψή μου στο συνδυασμό αυτό, βρίσκουμε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τριπλό φαινόμενο μόχλευσης. Μία πολιτική μόχλευση, μία τεχνική μόχλευση και μία χρηματοπιστωτική. Καταρχάς, στο πολιτικό επίπεδο, πέραν του ότι κάθε φορά που υπάρχει μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δημιουργείται εντύπωση ότι είναι παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να διαβάσετε τις εφημερίδες και τον τύπο στις ε, χώρες όπου επεμβαίνουμε, γράφεται ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που υποστηρίζει το ένα το άλλο έργο. Πέρα από το ζήτημα λοιπόν αυτό της προβολής, Υπάρχει και το ακόλουθο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό όργανο το οποίο νομίμως μπορεί να στηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ονομάζω μονοπόλιο των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο σε πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι κοινοτικά έργα τα οποία είχαμε προτιμάσει σε συνεργασία με τους, Ευρωπαϊ... με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξης, ξέρετε ότι μαζί έχουμε συγχρηματοδοτήσει πάνω από 100 έργα για ένα συνολικό ποσό 14 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, έχουμε μία πολύ καλή εμπειρία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη. Ορισμένες όμως φορές τα έργα τα οποία είχαμε προτιμάσει μαζί δεν καταφέραμε να τα χρηματοδοτήσουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε όχι δεν είναι δυνατόν αντιτίθεται στην κοινωτική πολιτική αυτό το οποίο κάνετε. Και αυτό για παράδειγμα συνέβη στη χρηματοδότηση αεροδρομίων στη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε όχι δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσετε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με την Ρωσία όσον αφορά τα δικαιώματα της ενέργειας κυκλοφορία, τα τέλη ενέργειας κυκλοφορίας, ενώ εμείς ουσιαστικά ήμασταν έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε το, σχέδιο αυτό, το έργο αυτό. Είμαστε ουσιαστικά το μόνο χρηματοπιστωτικό όργανο το οποίο πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα, τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε και η μόνη χρηματοπιστωτική υπηρεσία, ο μόνος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος υποχρεούται να έχει πρώτα την θετική γνώμη, τη σύμφωνη γνώμη και του κράτους μέλους το επιπεμβαίνει, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάνει μία διοργανική διαβούλευση και μάλιστα οποιαδήποτε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να εκφράσει την απόψή της και μερικές φορές έχουμε τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ή τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας ή τη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον που αντιτίθενται στο ένα ή στο άλλο έργο μας. Επομένω, είμαστε, είμαστε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ιδιαίτερα μοναδικό και ιδιαίτερο, γιατί είμαστε ο μόνο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο οποίο υπόκειται κατά αυτόν τον τρόπο στου κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ο μόνο οργανισμό, ο οποίο υπόκειται στι ε, γνωματεύσει ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα στο άρθρο 287 προβλέπεται ένας έλεγχος τριμερής Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε λοιπόν ένα μέσο, ένας μηχανισμός που έχει ως στόχο να στηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά τώρα το τεχνικό επίπεδο στο οποίο αναφέρθηκα, τεχνική διάσταση. Υπάρχει ένα επίπεδο αλληλοσυμπλήρωση ανάμεσα στην εμπειρογνωμοσύνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τα μακροοικονομικά στοιχεία, τα τομεακά στοιχεία, την πολιτική διάσταση ορισμένων έργων στι χώρε αυτέ, στι οποίε επεμβαίνει. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μια πολύ καλή πείρα όσον αφορά την τεχνική ανάλυση των σχεδίων των έργων. Θα μπορούσα να σα δώσω πάρα πολλά παραδείγματα. Θα αναφερθώ σε τρεις τομείς εφόσον ε, στην ε, μελέτη σας αναφέρεστε στην προστιθέμενη αξία της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αναφερθώ στην ενεργειακή απόδοση, το νερό και βλέπουμε ότι στους τομείς αυτούς όντως αναγνωρίζεται η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πολύ συχνά καλούνται οι δικές μας υπηρεσίες να τοποθετηθούν, να δώσουν εμπειρογνωμοσύνη για σχέδια τα οποία εμείς δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ούτως ή άλλως, γιατί η εντολή ούτως ή άλλως είναι εξωτερική. Για παράδειγμα στην Τουρκία χρηματοδοτήσαμε ένα αιωλικό πάρκο 135 ΜΒ με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και με κοινή συμφωνία ανάμεσα στις δύο τράπεζες είναι η δική μας τράπεζα η οποία προτίμασε όλο το σχέδιο πυρογνωμοσύνης. Έχουμε και το μνημόνιο συνεννόησης το οποίο υπεγράφει ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάμεσα στις δύο τράπεζες, όπου προβλέπεται ότι κάθε φορά που υπάρχει μία συγχρηματοδότηση θα πρέπει να διορίζουμε το θεσμικό αυτό όργανο το οποίο θα έχει την ηγετική θέση για τη διαχείριση του έργου και το όργανο εκείνο το οποίο θα ασχοληθεί με τη χρηματοδότηση. Δεν θα ήθελα να σας δώσω περισσότερα παραδείγματα αυτή τη στιγμή, πάντως υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε πάρα πολλού τομεί έχει αναγνωρισμένη γνωμοσύνη η οποία αλληλοσυμπληρώνεται με την εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να φερθώ τέλο και στην χρηματοπιστωτική διάσταση. Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι με το ίδιο ποσό από τον προπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να στηρίξει ένα πολύ σημαντικότερο τμήμα επενδύσεων. Αυτό εννοώ όταν αναφέρομαι στο φαινόμενο της μόχλευσης. Να αναφερθώ για παράδειγμα στο μηχανισμό χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων όσον αφορά την έρευνα. Αν δούμε πως είχε κατάσταση πέρυσι, είδαμε ότι χρησιμοποιήσαμε 390 εκατομμύρια από τον κοινοτικό προπολογισμό 772 εκατομμύρια από το κεφάλαιο της τράπεζάς μας και καταφέραμε να δώσουμε δάνεια για ερευνητικά προγράμματα για 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρηματοδότησαν σαστικά προγράμματα στο οποίο ιδιωτικό τομέα συμμετείχε με 16 δισεκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα 90% από τον κοινοτικό προπολογισμό δημιούργησε επιπλέον, επέφερε, προσέλκυσε από τον ιδιωτικό τομέα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρησιμοποιώντα πόρου από τον κοινοτικό προπολογισμό μπορούμε να προσελκύσουμε όλο και μεγαλύτερα ποσά. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ένα μονοπόλιο όσον αφορά τι υποχρεώσει τη. Σε καμία περίπτωση όμω δεν θέλει να έχει μονοπόλιο στην πρόσβαση του κοινοτικού προπολογισμού. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα προ αυτό. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο οργανισμό εκείνο ο οποίο βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για να προσελκύσει άλλου πόρου χρηματοδότηση κοινοτικών έργων από το δημόσιο και κοινοτικό τομέα. Ήμουνα στο Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα, ήμουνα σε επαφή με την επικεφαλή του Ταμείου Παρακαταθήκων, ο οποίο μου είπε, καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο εύκολο για μας να αποδεχθούμε να προσχωρήσουμε σε μια κοινή πρωτοβουλία αν, αυτό βρίσκεται, αν αυτή βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση με πρωτοβουλίες που θα αναλάμβαναν άλλα κράτη-μέλη. Αυτό κάναμε και με το σχέδιο Μαργκερίτ, όπου συνεργαζόμαστε με το Ταμείο Παρακατεθικών της Γαλλίας, με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς από την Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία είναι πολύ πιο εύκολο για όλους αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, να συνεργάζονται για τη χρηματοδότηση κοινοτικών έργων όταν εμπλέκεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όταν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι η προσέλγηση αυτών των επιπλέον πόρων θα είναι ιδιαίτερα αποφελή για τον κοινοτικό προπολογισμό. Θα πρέπει όμω να υπάρχει η εξή σημαντική προπόθεση. Ένα πάρα πολύ καλό έλεγχο, η κατάλληλη εποπτεία. Ο κύριο Καλβί το είπε πολύ καλά. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να συνάπτουμε συμφωνίε συμφωνίες, μνημόνια συνεννόησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να τελεί τον, ε, να επιτελεί το ρόλο αυτό τον εποπτικό τον οποίο έχει. Ενδεχομένως να προβλέπονται όμως και κάποιες κρυφές δαπάνες όσον αφορά τους μηχανισμούς αυτούς, αυτές τις διαδικασίες. Όντως θέλαμε να δούμε ποια είναι τα τέλη για την διαχείριση. Ποιε είναι οι προμήθειε, τι οποίε ενδεχομένω θα μπορούσε να έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την προσέλκυση αυτών των επιπλέον πόρων. Για την περίοδο 2007-2010 αν πάρουμε υπόψη μας όλες τις προμήθειες, εμείς λάβαμε 62 εκατομμύρια ευρώ από τον κοινοτικό προπολογισμό, εκ των οποίων τα 14 εκατομμύρια με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών όσον αφορά την χρησιμοποίηση των διαφορετικών ταμείων στο πλαίσιο του Τζέρεμι και του Τζέσικα. 62 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ ως προμήθειες για την περίοδο 2007-2010 το συνολικό ποσό των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τον κοινοτικό προπολογισμό στην τράπεζά μας είναι 4 ευρώ, 4,68 δις ευρώ. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, το επίπεδο προμηθειών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό το οποίο κοστολογούν οι ιδιωτικές τράπεζες και θα πρέπει να αφαιρέσετε από το ποσό αυτό όλα αυτά τα χρηματοπιστωτικά ωφέλη, τα reflows, τα οποία επιστρέφουν στον κοινοτικό προπολογισμό με τη μορφή απόδοσης όσον αφορά τις επενδύσει που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, για όλες τις ενέργειές μας στην ε, Μεσόγειο, τα reef έχουν φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ και θα φτάσουν τα 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ στα τέλη του έτους. Βλέπετε λοιπόν ότι και για το ζήτημα αυτό, να σας πω ότι όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία προφανώς Μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε εσείς, μπορεί η Επιτροπή σας να το κάνει αυτό. Θα ήταν ε, ενδιαφέρον λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο για τον κοινοτικό προπολογισμό. Όσον αφορά τώρα την κοινοτική εγγύηση, πρέπει να σας πω ότι η εγγύηση αυτή για τον κοινοτικό προπολογισμό ισχύει μόνο για τις ε, ενέργειες ε, αυτές οι οποίες γίνονται συγκεκριμένη εντολή 7-8% των δραστηριοτήτων μας ουσιαστικά δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν στην κοινοτική εγγύηση, ακόμα και για δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνουμε εμεί τον κίνδυνο χωρίς να ζητήσουμε την κάλυψη από τον κοινοτικό προπολογισμό. Για παράδειγμα, για τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες ε, χώρες 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ εμείς θα τους δώσουμε ως δάνειο μέχρι το 2013 λαμβάνοντας εμείς μόνοι μας τον κίνδυνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλύπτει αυτό ένα περιορισμένο μέρος των δραστηριοτήτων μας όλοι οι εμπορικοί κίνδυνοι αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό επιχείρημα είναι ότι στο παρελθόν δεν είχαμε ποτέ κανένα κίνδυνο για το κοινοτικό προπολογισμό, καμιά, καμιά απειλή από τότε που δημιουργήθηκε το Ταμείο Εγγύησεων δύο φορές μόνο το χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τη δεκαετία του 1990 για κάποια δάνεια που δόθηκαν στην πρώην Γιουκοσλαβία για ένα συνολικό ποσό 115 εκατομμύριων ευρώ και το ποσό το οποίο καλύφθηκε και επέστρεψε στο Ταμείο γησεων ήταν 204 ε, εκατομμύρια ευρώ και το 2003-2004 δόθηκε ένα δάνειο στην Αργεντινή, ένα συνολικό ποσό 9 εκατομμυρίων και το ποσό αυτό καλύφθηκε πάλι στη συνέχεια. Όλη η εμπειρία λοιπόν μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε κανένα επιπλέον κόστος από τον κοινοτικό προπολογισμό από τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου η κάλυψη ήταν περιορισμένη τους άλλως. Πιστεύω λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ότι υπάρχουν σαφή ωφέλη από το συνδυασμό του κοινοτικού προπολογισμού και των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θετικά στοιχεία τεχνικά, πολιτικά, χρηματοπιστωτικά, αρκεί βέβαια ο έλεγχος να είναι κατά τέτοιον τρόπο οργανωμένος, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη όσον αφορά τη χρήση των μέσων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάλστατ. Ήταν ε, πολύ εμπεριστατωμένη η παρουσίαση, σας, πολύ διεξοδική η παρουσίαση και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιπρόεδρο κύριο Φίσερ της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης να κάνει τη δική του δήλωση. Αλλά θα ήθελα να τον ε, παρακαλέσω να είναι πιο σύντομος από τον κύριο Μάλστατ. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε να είμαι ή δυνατόν σύντομος. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και ανασυγκρότηση και να σχολιάσω την μελέτη που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Επίσης, θα ήθελα να, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όσοι προσπαθήσαμε με αυτή τη μελέτη για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εργασία που έκαναν. Ε, δεν πρόκειται εδώ για μονόδρομο, όπως συνήθως ε, συμβαίνει ε, στους, ακαδημα, ακαδημαϊκούς όπου μιλάνε με αφηρημένους όρους. Εκείνοι ε, βασίστηκαν σε συνεντεύξεις και μίλησαν με εκπροσώπους των διαφόρων θεσμικών οργάνων και ε, θεωρώ ότι βασίστηκε η μελέτη αυτή σε μια πραγματικά διαλογική προσέγγιση. Η μελέτη αντανακλά την ανάγκη εκ μέρους, την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη σημασία της ε, συγχρηματοδότησης καθώς και τις αυξανόμενες σημασίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης και των σχέσεων μεταξύ τους. Η μελέτη το αναγνωρίζει αυτό πολύ ξεκάθαρα και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μήνυμα που εκπέμπει αυτή η μελέτη ε, λένε ότι υπάρχει μια επιθυμία διεύρυνση τη χρηματοδότηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση ω μέρο τη διαδικασία 2020. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση εκτιμά ιδιαίτερα στην ανάλυση του δικού μας οργανισμού και θεωρώ ότι καλύπτει τα τα βασικά στοιχεία του, του μοντέλου που λειτουργούμε βάσει το οποίο λειτουργούμε. Έχουμε την ε, ε, δυνατότητα να συμμετάσχουμε τώρα στην συγχρηματοδότηση. Είναι αλήθεια ότι η μόχλευση εδώ είναι πολύ υψηλότερη ορισμένες φορές επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη έχουν 63% των μεριδίων της τράπεζας και τέλος, όπως αναφέρει η μελέτη σας, εμείς ε, κάνουμε προσπάθειες αύξησης της ε, προβολής μας, του ρόλου μας στις ε, Βρυξέλλες. Και έχουμε έναν ειδικό εκπρόσωπο, την κυρία Μαντιπάν, η οποία κάθεται εδώ εξ ε, και είναι η δική μας εκπρόσωπος στις Βρυξέλλες. Χαιρετίζουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης όσον αφορά την πλατιά συνένεση για τις βασικές αρχές της συγχρηματοδότησης. Και θα ήθελα να αναφέρω τρεις αριθμούς που πραγματικά είναι ενδεικτικοί. Από την ε, αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης καθώς και 478 ε, δις ε, για ταμεία τεχνικής συνεργασίας. Και με τον τρόπο αυτό ε, καλύφθηκαν σημαντικά προγράμματα. Αυτή η συνεργασία ε, βασίστηκε στην, ε, κατέληξε στην θέσπιση τριών νέων εργαλείων. Η έκθεση βέβαια τονίζει κάποιες δυνατότητες ε, βελτίωσης όσον αφορά τα εργαλεία αυτά, τα μέσα αυτά, ε, στο πλαίσιο της ε, μελλοντικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας που βρίσκεται υπό εξέλιξη όσον αφορά τη βελτίωση για το μέγεθος των τραπεζών και εδώ συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση για την Επιτροπή όσον αφορά τους μηχανισμούς αναφοράς, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο στο επίπεδο των προγραμμάτων όσον και όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία και την ε, παροχή δεδομένων. Τα περιφερειακά μας γραφεία βρίσκονται επίσης σε επαφή με τις σημαντικές αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ε, προβολή ε, στην πράξη. Ε, η αξιολόγηση ότι η συγχρηματοδότηση είναι το πιο ενδεδειγμένο εργαλείο για την ανάπτυξη των αγορών μας βρίσκει σύμφωνος. Η συγχρηματοδότηση βασίζεται στην παράδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, και αυτό είναι ε, πιο σημαντικό στις χώρες εκείνης που είναι σημαντικό να γίνει πιο συνετή ε, διαχείριση των ε, ταμείων μέσω των ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων επιμερισμού του κινδύνου και χρηματοοικονομικής συνδρομής. Όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις του Προέδρου, τα όσα ανέφερε και τόσο είπε στη δική του παρέμβαση ότι όχι μόνο υπάρχει αυτό το υπόμνημα ε, ε, συνεννόησης, το μνημόνιο συνεννόησης το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μνημόνιο το οποίο παίρνουμε απολύτως σεβαρά αλλά επίσης θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας είναι το γεγονός ότι κάθε μέρα υπάρχει μια πολύ πρακτική συνεργασία όχι μόνο στο επίπεδο της έδρας των θεσμικών οργάνων αλλά στην καθημερινή μας ε, πρακτική δουλειά. Και εδώ ο Πρόεδρος ανέφερε ε, κάποια παραδείγματα όσον αφορά αυτή την εξαιρετικά καρποφόρα και αποτελεσματική συνεργασία. Δεν υπάρχει λοιπόν ανταγωνισμός και αλληλεπικάλυψη, αλλά αποτελεσματική συνεργασία που θα εξελιχθεί και στο μέλλον και θεωρώ ότι αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο απορρέει και από τους δύο οργανισμούς. Τώρα, ε, υπάρχει μία σύσταση η οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί κάπως παραπάνω, γιατί χρειάζεται να γίνει μια προσεκτική νομική αξιολόγηση. Αφορά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Από την άλλη υποστηρίζουμε πλήρως την ενδυνάμωση του συστήματος αναφοράς λογοδοσίας, το οποίο οδηγεί στην αύξηση της προβολής και ορατότητας, στην αύξηση της διαφάνειας, και την ε, βελτίωση των μηχανισμών λογοδοσίας των σημαντικών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και πάλι σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ και ε, ευχαριστούμε, ε, σας ευχαριστούμε και για τη μελέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Τόμας συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δώσατε τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος στη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και τους συμβούλους για την πολύ ακριβή στην έκφρασή της έκθεση. Η Γενική Διεύθυνση Εκφήν είναι υπεύθυνη για τις εγγύησει και όλες τις υποχρεώσεις του προπολογισμού. Το θέμα λοιπόν λογοδοσίας δημοσιονομικής και δημοσιονομικού ελέγχου γίνονται ακόμη πιο σημαντικά. Αλλιώ θα επέτρεπε στα προβλήματα να διαιωνίζονται. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε τις βάσεις ενός συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου και λογοδοσίας ώστε να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε τη χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων στο μέλλον. Σε αυτή την πτυχή της έκθεσης ήθελα να επικεντρωθώ ότι κάποια ζητήματα που εγείρουν οι συντάκτες της μελέτης ως προς τη χρήση των δημοσιονομικών εργαλείων γενικώ λόγου χάρη να οδηγούν στο σχόλιο ότι σε σύγκριση με άλλα εργαλεία πρέπει να πούμε ότι το καθοριστικό κριτήριο είναι οι, οι πολιτικές χώρο τη πολιτική. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί στόχοι χρηματοδοτήσιμοι από τη μια ή την άλλη τράπεζα. Άλλοι αρμόζουν περισσότερο από κάποιου άλλου. Τώρα, εάν κάποιος ε, παρεμβαίνει μέσω επιδοτήσεων, αυτό σημαίνει ότι έρχεται να διορθώσει τις αποτυχίες ε, της αγοράς. Όταν όμως κανείς ανατρέχει στη σηματοδότηση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει εταιρική σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και ανασυγκρότηση ή με άλλους ε, εταίρους τραπεζικούς και μη για να καλύψει τα κενά της αγοράς ακούσαμε ότι ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης είναι ίσως καλύτερος, διότι μέσω των δημοσιονομικών εργαλείων ουσιαστικά αναγκάζουμε περισσότερους φορείς να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις αποτυχίες της αγοράς. Όπως σωστά είπαν οι συμβουλοί μα τελικώς, υπάρχει και ένα θέμα ισορροπία. Υπάρχει καλύτερος δημοσιονομικός έλεγχος όταν υπάρχουν ε, επιδοτήσεις και Σε ορισμένου πολιτικού τομεί τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν υπάρχει συνεργασία των θεσμικών οργάνων με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή την ισορροπία έχουμε αναζητήσει ως τώρα. Επίση, η έκθεση, η μελέτη μάλλον, θα μπορούσε να δει καλύτερα την δυναμική εξέλιξη κάποιων από τα εργαλεία χρηματοδότηση, όπω τον τομέα τη ανάπτυξη, τη καινοτομία, τη έρευνα, Εκεί έχουμε μακρά πείρα συνεργασία και εργασία με τέτοια δημοσιονομικά εργαλεία. Στα διευθυντικά ταμεία, Κάποιοι μηχανισμοί χρηματοδότηση είναι πιο καινούργοι. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά να τα δούμε με περισσότερη προσοχή. Το Τζέρεμι αναφέρθηκε στην παρουσίαση. Θα έλεγα ότι εδώ το ποτήρι μπορούμε να το δούμε και κατά ένα τρίτο γεμάτο, ε, αντί για δύο τρίτα άδειο. Θα ζητούσα λοιπόν από του συντάκτε τη μελέτη να δούνε και τον δυναμικό χαρακτήρα των ε, μέχρι σήμερα εξελίξεων και όχι μόνο από την θεωρητική, την ακαδημαϊκή την ε, άποψη. Κατά την εξέταση ζητημάτων όπως η διαφάνεια, η διακυβέρνηση, ζητήματα που ορθώς θέτουν οι ε, συμβουλή μας εδώ. Νομίζω ότι κατά την κίνησή μας προς τα μπρος θα πρέπει να διδαχθούμε από την ως σήμερα πείρα μας και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια όταν έχουμε να κάνουμε με δημοσιονομικά εργαλεία. Είμαι βεβαίω ότι σε άλλες ευκαιρίες συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή Ήδη έχετε δει κατά πόσο μπορεί να υπάρξει σταδιακή αύξηση της δημοσιονομικής ρικοδότησής μας στο μέλλον και έχω δει διάφορες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά εργαλεία στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη κοιτάζει πώς θα αντιμετωπιστούν οι πλατφόρμες του χρέους και των αξιογράφων στο μέλλον ε, ώστε να μπορεί να υπάρχει σωστή αξιολόγηση του κινδύνου, αξιολόγηση της ε, του πώς συνδυάζονται μεταξύ των διάφορα δημοσιονομικά εργαλεία. Οι συντάκτες λοιπόν της μελέτης μπορούν να έχουν μια πιο διορατική ματιά. Χρειαζόμαστε μια καλύτερα προετοιμασμένη βάση κανόνων για τα δημοσιονομικά εργαλεία. Αντί λοιπόν να βλέπουμε μόνο τα κενά και τις ελλείψεις που μπορεί να έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία, καλό είναι να σκεφτούμε και στην πράξη και να σκεφτούμε πώς μπορούμε στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Τέλος, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο το οποίο καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη ε, και σε σχέση με τη μελέτη. Όταν τα σημερινά δημοσιονομικά εργαλεία σχεδιάστηκαν ε, στις αρχές αυτής της δημοσιονομικής περίοδου, κατά το 2007, βλέπουμε τα πράγματα από την σκοπιά την πολιτική για το πώ θα μπορούσαμε να βρούμε δημοσιονομικά εργαλεία που να αντικαθιστούν τι δωρεέ. Νομίζω όμω ότι η χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση των δημοσίων χρεών έχει ε, επιφορτήσει με ένα περαιτέρω βάρο ε, τη λειτουργία των εργαλείων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Τράπεζα Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση, ιδίω η δεύτερη, έχουν διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην σωστή εφαρμογή των εργαλείων όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί, αλλά και στο να παράσχει πιστός και, αξιο... και ασφάλεια στην ευρωπαϊκή οικονομία καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Έτσι λοιπόν προσθέθηκαν νέοι πολιτικοί στόχοι σε, όλο, σε όλη τη σύλληψή μας των δημοσιονομικών εργαλείων ε, αναγκαστικά λόγω της κρίσης. Τέλος, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως ε, ο κ. τα είπε σωστά, και την ελέγχουμε και πρέπει να, βλέπουμε, να επαληθεύουμε το κάθε πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν έχουμε και μια συμμετοχή του 3%, οπότε προσπαθούμε να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές μέσω της διακυβέρνησης ακόμη και με πολύ λιγότερα, ακόμη και αν έχουμε λιγότερα δικαιώματα ως, ε, από το καταστατικό της τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να προάγουμε την καλή λειτουργία και αυτών των θεσμικών οργάνων και όλων γενικώ των θεσμικών οργάνων, δημοσίων και μη. Ε, Σημειώνω το σχόλιο ότι μέσω τη διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών και θεσμικών οργάνων θα πρέπει να προάγουμε την καλή διακυβέρνηση. Θα σταματήσω εδώ για την ώρα για να μην εξαντλήσω το χρόνο και είμαι διαθέσιμο για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα έχουμε πλέον μια πληθώρα πληροφοριών και ε, υπάρχουν και κάποιες ε, διχογνωμίες σε σχέση με τα όσα ακούσαμε. Υπάρχει ένα μικρός μάλλον κατάλογος ομιλητών. Ο Λάιος Όκρους και μετά η Γκρέσλε. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω αυτή τη στιγμή τους uh, συντάκτες των ε, μελετών αυτών, της μελέτης αυτής. Θα ήθελα να ζητήσω όμως από τους ε, συντάκτες της ε, μελέτης στην επόμενη φάση της μελέτης και βέβαια ξέρω ότι δεν εξαρτάται τόσο από αυτούς, εξαρτάται, τόσο από, εξαρτάται περισσότερο από εμά. εμείς πρέπει να θέσουμε το αίτημα. Θα ήθελα λοιπόν να εντάξουν στο πεδίο της μελέτης αυτής το ακόλουθο. Ποιες θα είναι οι επιπτώσει τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη για τον κοινοτικό προπολογισμό. Είναι πολύ συγκεκριμένη ουσιαστικά η ερώτηση. Στην δημόσια πολιτική, όπως γνωρίζετε, γίνεται μια πολύ ισχυρή διάκριση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την επίτευξη αποτελεσμάτων. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε περισσότερο στην διαδικασία, αν είναι όντω γρήγορη, αν μπορεί να θεσπιστεί ένα έργο γρήγορα, αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με τρόπο ευέλικτο και γρήγορο. Και όσον αφορά την επίτευξη έπειτα των αποτελεσμάτων, αναφερόμαστε περισσότερο στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το έργο αυτό. Δυστυχώς, όταν συζητάμε επιπτώσεις για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ουσιαστικά μία λεπτή ισορροπία την οποία πρέπει να διατηρήσουμε. Και θα ήθελα εδώ πέρα να είχα την γνώμη των συντακτών της έκθεσης. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη δημόσια πολιτική που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν αλλοιούμε συγκεκριμένα έργα, βλέπουμε ότι Όσο μικρότερο είναι ο κίνδυνο για τον κοινοτικό προπολογισμό, τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνο για τι χώρε. Βέβαια, ξέρετε ότι πολλά έργα έχουν μία εγγύηση εθνική και ότι ε, τα... όταν, όταν μάλλον κάτι δεν πηγαίνει καλά στη συνέχεια μπορούν τα κράτη μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη που έχουν αναλάβει την εθνική αυτή ευθύνη για να αποπληρώσουν κάποια δάνεια σε περίπτωση πτωχεύσεων για παράδειγμα. Σε ορισμένες ε, χώρες έχουμε δει να, γίνεται το παράδειγμα, να, να υλοποιείται το παράδειγμα. Αυτό το είχα δει και στο προηγούμενο πόστο το οποίο είχα και στο οποίο είχα μείνει για 8 χρόνια. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπε ο κύριος Μέιστατ. ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα, χρησιμοποιεί, θα χρηματοδοτεί όλο και περισσότερα έργα όπου δεν θα υπάρχει μια εγγύηση από τα κράτη αυτά καθ' αυτά, όπου το 80% του κινδύνου ουσιαστικά θα τον λαμβάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος θα είναι μεγαλύτερος για τον κοινωνικό προπολογισμό. Αυτό το ζήτημα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να λύσουμε περισσότερο και αν πιέσουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης προς τον δρόμο αυτό θα πρέπει να γίνουν και απαραίτητε αναλύσεις. Να δούμε δηλαδή ποιε ήταν οι επιπτώσει από μια τέτοια ανάμειξη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη και ποιε ήταν επιπτώσει στον κοινοτικό προπολογισμό. Θα ήθελα λοιπόν επ' αυτού να είχα την άποψη των συντακτών τη μελέτη. Γιατί πολύ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να δουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερα σύγχρονα μέσα στη χρηματοδότηση. αλλά το ζήτημα πάντα είναι πώς θα καταφέρουμε να επιμερίσουμε διαφορετικό τρόπο το κίνδυνο. Και όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε μέσα στη χρηματοδότηση, υπάρχουν όλο και περισσότεροι κίνδυνοι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο πρέπει να κατανεμηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ίγκε έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η μελέτη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και είναι η πρώτη μελέτη η οποία πραγματικά ασχολείται με το θέμα αυτό της χρησιμοποίησης των ε, μέσων αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στο δημοσιονομικό κανονισμό, γιατί εκεί παίζουν σημαντικό ρόλο αυτά τα εργαλεία. Ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης ε, μας παρουσίασαν αυτά τα εργαλεία. Μόνο που τώρα βρισκόμαστε πρώτου επόμενου βήματος, η διεύρυνση της αξιοποίησης των εργαλείων αυτών μέσω ιδιωτικών τραπεζών το σχέδιο του δημοσιονομικού κανονισμού ήδη προβλέπει τα επόμενα βήματα και θα ήθελα να σα το επισημάνω γιατί έχουμε καταθέσει εδώ σχετικές τροπολογίες. Είπαμε για παράδειγμα ότι αυτό το οποίο ε, θα θέλαμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και είπαμε ότι θα θέλαμε να έχουμε ένα έγγραφο εργασία. Ε, στα όσα λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, το πώς χρησιμοποιούνται, ποια είναι τα αποτελέσματα και τι γίνεται με το θέμα του κινδύνου, το οποίο πράγματι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό το οποίο λέει η μελέτη για τα προβλήματα του ελέγχου του προπολογισμού και το θέμα κατά πόσο πετυχαίνουμε τους στόχους μας μέσω αυτών των εργαλείων ή των μέσων, ε, είναι σημαντικό. Ε, το ζήτημα Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση. Ε, ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση ε, ορισμένων προγραμμάτων και νομιμοποιείται χρήση του, αλλά θα με ενδιαφέρε να μας πούν οι συντάκτες της μελέτης κατά πόσο έχουν ενδείξεις για τις ελλείψεις όσον αφορά την καθοδήγηση αυτών των, ε, τη χρησιμοποίηση αυτών των εργαλείων γιατί πάνω από 50% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελικά ε, δεν κατευθύνονται σε αυτά τα εργαλεία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα των ευρωομολόγων, δηλαδή ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να θεσπίσουμε για τα ευρωομόλογα. Και θα ήταν ε, σημαντικό οι συντάκτες εφόσον κάνουν ένα follow-up να μας πούν ποια είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα ήθελαν οι ίδιοι να μας προτείνουν. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, Ιζαμπέλ φαίνεται ότι έχει καλυφθεί ή όχι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μπόρεσα να παρακολουθήσω αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Δεν έχω καταφέρει ακόμα να διαβάσω ολόκληρη τη μελέτη, αλλά πρέπει να πω τα εξή. Από τη μια συνοπτικά η έκθεση επιστά την προσοχή σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα διαφάνειας το Κόστο τη διακυβέρνηση, τη σημασία του ελέγχου. Ακούσαμε εδώ κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τη ίδια, ότι θέλει να κάνει περισσότερα και να μας δώσει και πρόσθετα στοιχεία, αλλά από την άλλη μόλι συζητήσαμε και την έκθεση τη Κυρία Γκρέσλε. Παρομοίω και εκείνη μας επεσήμανε με όλες τις τροπολογίε την ανάγκη απλούστευση. Με διαφόρων πολύπλοκων ε, διαδικασιών. Βλέπουμε λοιπόν από τη μια τον κλασικό ευρωπαϊκό προπολογισμό και τη διοργάνωσή του, από την άλλη την περιπλοκότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που συμμετέχει σε μια σειρά ποικίλων προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι η πολυπλοκότητα υπάρχει παντού, ακόμη και στον ίδιο τον προπολογισμό μας. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε να αναζητήσουμε τις λεπτομέρειες και τις διορθώσεις που χρειάζονται στον ίδιο μας τον προπολογισμό. Εδώ λοιπόν το θέμα είναι κατά πόσον υπάρχει επιστροφή των δανείων μεν, αλλά και από την ιστορία μέχρι τώρα που έχετε, το ιστορικό σας, την πείρα σας, βλέπουμε ότι κατά τρόπο θεαματικό δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ε, είδαμε τους αριθμούς, τα αριθμητικά στοιχεία. Οι ευρωπαϊκές εγγύσεις είναι το 7% των συναλλαγών, ιδίω αυτών που κατ' εντολή ε, Δεν βλέπω λοιπόν αυτή η απειλή να είναι τεράστια, έναν ε, δεν τιμήσει τις υποχρεώσεις του είναι περιορισμένη η απειλή. Στην πράξη ως τώρα δεν υπήρξε κίνδυνος, ε, σοβαρή απειλή για τον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο μου παρατηρήσεις, με την επιφύλαξη βεβαίως ότι θα μελετήσω εντελεχώς τη μελέτη και τις απαντήσεις που μας έδωσαν οι δύο Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Okay, wir haben jetzt... Ωραία λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε μια πραγματικά μακρά διεξοδική συζήτηση και οι δυο μας επιστήμονες άκουσαν ε, ποια είναι τα επιπλέον ε, αιτήματά μας που δεν ε, ικανοποιούν μέχρι στιγμής οι μελέτες. Ο Εβάλο Κάλφιν θα μας ε, επισημάνει τώρα μια δυνατότητα διεξόδου ε, το πώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε ενδεχομένω τη συνεργασία εδώ σε αυτό το σημείο. much, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ως προς τους συντάκτες της μελέτης να υπογραμμίσω τρία στοιχεία απευθυνόμενος εκείνος. Πρώτα απ' όλα ότι προφανώς η μελέτη επισημάνει, επισημάνει ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι τα πορίσματα της έκθεσης θα συμμερίζονται όλα τα θεσμικά όργανα ή το κοινοβούλιο. Σίγουρα, ε, ο στόχο είναι βέβαια να ξεκινήσει εδώ μια ουσιαστική συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Έχουμε διαφορετικέ απόψει και αυτή είναι και η δουλειά μα. Αυτό διευκολύνει το έργο μας και είναι και απόψει μας ε, πιο θεμελιωμένες όταν λαμβάνουμε αποφάσεις. Έπειτα, κάποια αποτελέσματα που που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο δικό μας έργο και εμείς στην Επιτροπή μας. Πρώτον, συμφωνούμε ότι η συγχρηματοδότηση με την ως τώρα πείρα μας είναι θετική ε, διαδικασία. Ω προ τα εργαλεία που ω τώρα έχουν χρησιμοποιηθεί, τα νέα που έχουν αναπτυχθεί μετά την οικονομική κρίση και τα αναφέραμε πολλά από αυτά. Πολλά τα ετοίμασε η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλε αυτέ οι εμπειρίες ω τώρα ήταν θετικέ. Έπειτα βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα και ανάγκη να αναζητήσουμε βελτιώσει στου υπάρχοντε μηχανισμού Στην έκθεση έχουμε να κάνουμε με ζητήματα διαφάνεια, προβολή ελέγχου Χαίρομαι πάρα πολύ που και οι δύο ευρωπαϊκές τράπεζες είναι έτοιμες να εργαστούν για τα ζητήματα αυτά, για να τα αντιμετωπίσουν. Και αυτό θα το έχουμε κατά νου στην συνέχεια της συζήτησης για όλα αυτά. Κατά τρίτον, υπάρχει δυνατότητα να επεκταθεί περαιτέρω η συγχρηματοδότηση. Όπω είπε και ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή, βεβαίω θα πρέπει πολύ προσεκτικά να αποφασίσουμε για ποιου πολιτικού τομεί. Προφανώ όχι σε όλου του Ευρωπαϊ... τομεί ευρωπαϊκή πολιτική ε, δεν γίνεται να ανατρέξουμε στη συγχρηματοδότηση, αλλά θα έπρεπε να αναζητήσουμε τα καταλληλότερα εργαλεία για κάθε περίπτωση. Το να προσπαθούμε λοιπόν του υπάρχοντες μηχανισμού να του βελτιώσουμε, τους βελτιώσουμε και να σκεφτόμαστε ήδη ποια νέα εργαλεία μπορεί να μα διευκολύνουν στο μέλλον είναι κάτι που είναι χρήσιμο. Βεβαίω, μιλώντα για τα επιπλέον εργαλεία, και με αυτό θα θέλω να ολοκληρώσω, καλό είναι να έχουμε υπόψη και τα επίπεδα κινδύνου. Κάτι που και ο Λάιος ανέφερε. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά βεβαίω. Άλλο ε, ο κίνδυνο τη τράπεζα και άλλο ο κίνδυνο των ε, κρατών, ε, των κυρίαρχων κρατών, των δικαιούχων των ίδιων. Όμως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια καλή άποψη της σωστόρα τώρα κατάστασης. Ξέρουμε ότι ε, η απειλή και ο κίνδυνος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Κάποιες ε, φορές σχεδόν μηδενικός. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι οι χώρε δικαιούχοι δεν αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο. Εκεί είναι αυξημένο ο κίνδυνο, μάλλον. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε τι επίπεδο κινδύνου μπορούμε να αναλάβουμε και σίγουρα θα θέλαμε να είναι στο δυνατόν πιο περιορισμένο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και ο σχεδιασμό νέων εργαλείων είναι ένα θέμα, θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειε, ήδη θα έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συντάκτες της μελέτης και τους ε, διευθυντές των δύο Ευρωπαϊκών Τραπεζών που παρουσίασαν τις δηλώσεις τους. Θα τα σκεφτούμε όλα αυτά πολύ σοβαρά στο έργο μας, στο μελλοντικό μας έργο στην Επιτροπή Προβλογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι έχουμε πολιτικούς στόχους και για την επίτευξη αυτών των, την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στόχων έχουμε διάφορα εργαλεία στη διάθεσή μας και προσπαθούμε να αναπτύξουμε και άλλα εργαλεία γιατί γι' αυτό άλλωστε ασχοληθήκαμε με τα να καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα ήδη φυστάμενα εργαλεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τους προβληματισμούς μας και μελλοντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Τουλάχιστον εμείς έχουμε τη βολή να το κάνουμε. Τώρα, για να μπορέσει να συνεχίσει να δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότηση, έχουμε και εμείς καταρτήσει μια γνωμοδότηση, Ιβάλλο, τη δική σου, την οποία ε, συζητήσαμε για την εγγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απόκτηση νέων μεριδίων στο τεμαχητοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης. Έχουν κατατεθεί εδώ δύο τροπολογίες και νομίζω ότι μπορούμε να τις ψηφίσουμε. Δεν χρειάζεται κατά την άποψή μου περαιτέρω συζήτηση. Υποθέτω ότι συμφωνείς. Έχουμε δύο τροπολογίες, καταρχήν για την ιδεολογική σκέψη 5α και για το άρθρο 1 δύο τροπολογίες του Μικελ Πόρτας και της Γιουν Κλούτε. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μπλοκ. Ωραία, δεν έχετε κάποια αντίρρηση. Λοιπόν, τις ψηφίσουμε από κοινού. Ποιος είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών. Τρεις ψήφοι. Ποιος είναι κατά των τροπολογιών αυτών. Ποιος απέχει. Λοιπόν, μια σημαντική πλειοψηφία κατά των τροπολογιών αυτών. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την έκθεση ως έχει. Υπέρ παρακαλώ. κατά αποχές ουδής. Λοιπόν, εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία, θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ όλους όσους ε, έλαβαν μέρος στον τελευταίο γύρο των συζητήσεων, τους συντάκτες μας, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, τον ε, διευθυντή της ΕΚΦΙΝ και όλους όσους ε, προσήλφαν εδώ, άκουσαν προσεκτικά τις συζητήσεις ή συμμετείχαν σε αυτές. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το πακέτο της Λισαβόνας. Ράιμερ, Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί μετά την τελευταία συνεδρίαση στις 13 και 14 Απριλίου που κάναμε μια σχετική συζήτηση δεν έχω να σας πω σήμερα κάτι καινούριο. Ε, θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι στις 15 και 16 Μαρτίου είχαμε μια εσωτερική συζήτηση στη βάση των συμπερασμάτων της νομικής μας υπηρεσίας και σημαντικό για τις ε, ομιλίες εδώ με το Συμβούλιο. Το γεγονός ότι αύριο θα συναντηθώ ε, με, την, ε, τον εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας για να δούμε πού είναι τα περιθώρια διαπραγματεύσεων και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικά της ψηφοφορίας ή όχι. Η φυστάμενη διοργανική ε, συμφωνία, εξακολουθεί να ισχύει. Μέχρι ότου έχουμε μια νέα διοργανική συμφωνία. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τα άρθρα τα οποία αντιβαίνουν στη συνθήκη. Δεύτερον, έχουμε τη δέσμευση, την υποχρέωση ε, σε μια συγκεκριμένη χρονική προθεσμία να δούμε κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι και βεβαίως ε, θα πρέπει ε, να γίνουν ε, οι διαπραγματεύσεις για το άρθρο 312 της συνθήκης παράγραφος 2 και θα πρέπει να σας καταστήσω σαφές ότι είναι θλιβερό το γεγονός ότι η πλευρά του Συμβουλίου προφανώς μέχρι σήμερα δεν έχει το κοινό ενδιαφέρον να επιτύχει μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο για το πώς θα πρέπει να οργανώνεται μελλοντικά η διαδικασία αυτή σύμφωνης ε, ε, γνώμης. Ε, και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί ο δεδομένο τρόπος να συμπεριληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ένα κείμενο προβληματισμού ε, της 25ης Τετάρτου με το κείμενο που είναι μια σύνοψη των όσων έγιναν. Ε, μου είπαν ότι στη σελίδα 3 στην πρώτη παράγραφο ε, υπάρχει μια κάπως περίεργη διατύπωση όσον αφορά τις αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες ε, πράγματι αναφέρονται στην υφιστάμενη ευελιξία για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού προγραμματισμού, δηλαδή την εφαρμογή του άρθρου 21-23 ε, στη βάση της νομικής ερμηνείας από την πλευρά του Συμβουλίου. Θα γίνει αυτή η προετοιμασία από την πλευρά του Συμβουλίου με τη διαφορά ότι το Contingency Reserve είναι κάτω από 0,03 του ΑΕΠ. Ελπίζω να κινητοποιηθεί το Συμβούλιο με μια ειδική πλειοψηφία με την ε, διαφορά ότι θα γίνει μια αναθεώρηση του 0,03% και θα αντισταθμιστεί από το Συμβούλιο με περιθώρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να πούμε ότι στο παρελθόν σε τέτοιου είδους αναθεωρήσεις ποτέ δεν ξεπεράσαμε το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά γνωρίζουμε ότι τα περιθώρια αυτά γίνονται όλο και πιο στενά και αυτό όχι μόνο από θεωρητική άποψη αλλά de facto τελικά οδηγούν σε ένα περιορισμό των δυνατοτήτων αναθεώρηση ή θα μπορούσαν να οδηγούν σε μια τέτοια συρρήκνωση των περιθωρίων για το μέλλον. Η συζήτηση στην τελευταία συνεδρία, συνεδρίαση κατέστησε σαφές ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ε, λογικές συζητήσεις, πραγματεύσεις με το Συμβούλιο εν σχέση και με πώς μπορούμε να οργανώσουμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλου το ζήτημα της ειδικής πλειοψηφίας και της ομοφωνίας και κατά πόσο υπάρχουν ενδεχομένω άλλες δυνατότητες μιας αντιστάθμισης μέσω ε, με εργαλείων ευελιξίας ή κάποιων άλλων ε, δυνατοτήτων. Ε, θα πρέπει να ζυγίσουμε όλα αυτά τα θέματα και θα ήθελα σήμερα απλώς ε, να πω ότι θα πρέπει να δω καταρχήν ποιο είναι το περιθώριο που έχει η Πρεδρία του Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κανονικές και σωστές διαπραγματεύσεις σε σχέση με τις αντισταθμίσεις τις οποίες προανέφερα, ενδεχομένως θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου η Επιτροπή Προπολογισμού θα πρέπει να δει κατά πόσο θα ολοκληρώσει με αρνητικό τρόπο αυτή τη διαδικασία σύμφωνη γνώμη. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν, ότι μπορούν να γίνουν κάποιε θετικέ διαπραγματεύσει. Οι σκιώδει και οι συντονιστέ ε, είχαν συναντηθεί πριν από την τελευταία συνεδρίαση και συζήτησαν και θα ήθελα να προτείνω υπό την έννοια της ε, σύσταση ομάδα εργασία 27 έω 30 Μαου, ενδεχομένω μεταξύ της ε, επιτροπή προπολογισμών και να έχουμε να κάνουμε μια ε, ε, συνεδρίαση και να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Εάν η πλευρά του Συμβουλίου δεν είναι διατεθειμένη να το πράξει, θα πρέπει να πάρουμε εμείς τη δική μας απόφαση. Αν ε, υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις, τότε θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις, εάν όχι, τότε εμείς με κάθε ηρεμία θα πάρουμε τη δική μας απόφαση σε, την, ε, σε αυτό το θέμα. Γιατί όπως είπε και η νομική υπηρεσία, ε, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε με αυτόν τον τρόπο την φωλιά μας και να βρεθούμε χαμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης θέλει να πάρει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ράιμερ, για αυτό το έγγραφο χασμού το οποίο μας έδωσες, περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση, τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα και κάνεις και κάποιες προτάσεις για άλλα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ευελιξία, που ουσιαστικά μας επαναφέρουν σε προηγούμενες θέσεις. Για την πολιτική μου ομάδα αυτό μπορώ να πω είναι ότι σε υποστηρίζουμε πλήρως. Ευχόμαστε καλή επιτυχία αύριο στις ε, συζητήσεις που θα έχεις. Ξέρουμε ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο και ότι ενδεχομένω ε, να πρέπει ε, όντως να τονίσουμε ότι με ιδιαίτερο σθένος υπερασπίζουμε τη θέση μας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για τις μελλοντικές συζητήσεις που θα γίνουν για το πολιετές πλαίσιο αλλά και γιατί όταν θα συζητήσουμε για τον κοινοτικό προπολογισμό 2012 θα πρέπει να επιλύσουμε τα εκεί υφιστάμενα προβλήματα. Και πιστεύω ότι τα δύο αυτά ζητήματα θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και στο μέλλον. Επομένως, δείξε δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά να μην παίζουμε με τη φωτιά όταν πρόκειται για τον προπολογισμό του 2012. Ράιμερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη, γιατί συζητήσαμε κατ' επανάληψη το θέμα αυτό και όπως έλεγε ο κύριος Μπέγκε, ε, δεν έχουμε ακόμα τις πρώτες πληροφορίες από τις συναντήσεις με το Συμβούλιο. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η θέση του Κοινοβουλίου αύριο στι συζητήσει με την Ουγγρική Προεδρία θα πρέπει να είναι απολύτω ξεκάθαρη. Και το είπε άλλωστε ξεκάθαρα, Ράιμερ είτε θα ανοίξουμε κάποιες αληθινές πραγματικές διαπραγματεύσεις γιατί μέχρι στιγμής ε, οι διαπραγματεύσεις βασίστηκαν σε κάποιες προτάσεις του Συμβουλίου που αγνοούσαν πλήρως τη θέση του Κοινοβουλίου. Ή αλλιώς ε, θα πούμε όχι, θα αρνηθούμε την πρόταση του Συμβουλίου. Αυτό θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εάν αυτοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν, τότε θα διαπραγματευτούμε και εμείς. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής και αυτό που αυτή τη στιγμή ισχύει η ειδική πλειοψηφία, τα θέματα ειδική πλειοψηφία, η, η ζητήματα Οργανική Οργανικής Συμφωνίας. Ε, αυτή είναι η βάση που έχουμε. Ε, και αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι μεγαλύτερη ευελιξία δεν ε, βασιζόμαστε στην πρόταση του Συμβουλίου. Βασιζόμαστε σε αυτό το οποίο έχει εγκριθεί. Το Συμβούλιο έχει τη δική του πρόταση και εμεί έχουμε τη δική μα ε, πρόταση. Και αν δεν είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε πραγματικέ αληθινέ διαπραγματεύσει, τότε εμεί θα αρνηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η Χέλγα Τρίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Ράιμερ για την παρουσίασή σου. Θα ήθελα να επανέλθω εν συντομία στο θέμα των πολιτικών συνεπειών. Και εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια κινητοποίηση στο Συμβούλιο και ε, να υπάρξει μια κίνηση στην, ε, στο επίπεδο της συζήτηση. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε η Επιτροπή δεν θα πρέπει να δεχτεί αυτό που επιθυμούν να μας επιβάλλουν. Και εμείς θα μείνουμε σε αυτό το οποίο από κοινού συμφωνηθέντα. Ε, Ράιμαρ, αυτό είναι σημαντικό, να υπάρχει καθαρότητα και να έχεις αυτή την ξεκάθαρη εντολή. Δηλαδή, είμαστε διατεθειμένοι για διαπραγμάτευση, αλλά εφόσον υπάρχει μια πολιτική μετατόπιση, βούλης πολιτικής μετατόπισης εκ μέρους του Συμβουλίου. Αλλιώς θα το κάνουμε. Ωραία λοιπόν, μετά από όλες αυτές τις δηλώσεις, λέει ο πρόεδρος, νομίζω ότι ο Ράιμερ θα είναι πολύ καλά εξοπλισμένος. Ε, εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και δεν το κάνει κάθε πολιτική ομάδα, να ορίσει το σκιώδη για αυτή την ομάδα εργασία. Ούτε στο Ράιμερ να γνωρίζει σε ποιον μπορεί να απευθυνθεί. Όταν ε, θέλει να δει ποιες είναι οι θέσεις των πολιτικών ομάδων. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε εδώ αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε, πόσο μακριά θα πάμε αυτή τη φορά, θα καταφέρουμε. Τώρα ε, έχουμε δύο, θα πρέπει να αφήσουμε δύο γνωμοδοτήσεις ε, δεν βλέπω την εισηγήτριά μας, αλλά την πρώην εισηγήτριά μας, η οποία πάντοτε είναι αρμόδια για την αλία. Δεν είναι εδώ. Ελγα, θα αναλάβει εκ μέρους της Αλφονσίν. Ε, θα πρέπει να σου πω, Γιούτα, ότι δεν είμαι προετοιμασμένη, παρκώς προετοιμασμένη. Ωραία, ίσως με τη βοήθεια του συνεργάτη του, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να κάνουμε την ψηφοφορία. Ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν έχουν ε, ε, περάσει καμιά τροποβολογία. Απλώς ε, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε σαν πρώην μέλος της Επιτροπής Αλίας να κάνεις κάποια δήλωση. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση για το πρωτόκολλο με τις Σεϊχέλες. Ε, Όποιο συμφωνεί παρακαλώ να υψώσει το χέρι. Κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Ωραία. Με μεγάλη πλειοψηφία γίνεται δεκτό. Τώρα είναι η συμφωνία με το Σαοτομέ και Πρίνσιπε υπέρ της γνωμοδότησης του εισηγητού κατά αποχές ωραία με, με την ίδια πλειοψηφία γίνεται δεκτό τώρα στην μεταφορά των ε, κονδυλίων για τη μεταφορά των ε, κονδυλίων που πρέπει, τη μεταφορά των πιστώσεων που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε να ε, πετύχουμε την προθεσμία της Τετάρτης Πέμπτου. Στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής αναβλήθηκε η ψηφοφορία αυτή για τη μεταφορά πιστώσεων, γιατί υπήρχαν κάποια θέματα διευκρίνηστα για την εισηγήτρια. Η εισηγήτρια δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα, αλλά βεβαίως έλαβε όλες τις ε, πληροφορίες που μας ε, έστειλε η Επιτροπή και τις, τις είδε λοιπόν, τις εξέτασε, τις μελέτησε και είναι τώρα υπέρ αυτής της μεταφοράς πιστώσεων. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πώς συμφωνείτε με τη σύσταση της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ της μεταφοράς πιστώσεων. Ευχαριστώ. Κατά, παρακαλώ. αποχές. Ωραία λοιπόν. Εγκρίνουμε λοιπόν τη μεταφορά πιστώσεων. Τώρα θα έρθουμε στο σημείο 12 Θα ήθελα να σε ρωτήσω σαν Ναι, εδώ ξέρω τι έχω να πω, Γιούτα. Αφόρ. Το ελεκτικό συνέδριο θέλει να δώσουμε έγκριση για το ST7 σε μια νέα γραμμή. Πρόκειται για μια πολιτική του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες ασφάλειας εσωτερικές πλέον του ελεκτικού συνεδρίου, οι οποίες θεωρούνται πολύ λιγότερο δαπανηρές από ό,τι να χρησιμοποιηθούν εξωτερικές ε, υπηρεσίες. Επομένως, προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ, καθότι η κίνηση αυτή είναι πολύ σωστή. Υπάρχουν παρεμβάσεις. Όχι, άρα μπορούμε να συμφωνήσουμε την πρόταση της σύστασης της υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, το 13 έχει αναβληθεί που αφορά την πολιτική ακινήτων. Και αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση Τώρα θα έρθουμε στην ΕΜΖΑ και την ΕΝΙΖΑ. Θα ξεκινήσουμε με την ΕΝΙΖΑ. Όπως ξέρουν οι συνάδελφοι, ήταν μια υπηρεσία για τα δίκτυα και την ε, ασφάλεια πληροφοριών ε, ούτως ώστε τα δίκτυα και πληροφορίες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ασφαλή. όταν αποφασίσαμε την Νίζα μέσω κανονισμού, ταυτόχρονα διαπιστώσαμε το τέλος της ΕΝΙΖΑ. Αλλά δεν ήρθε αυτό το τέλος. Ε, και θα θυμούνται οι συνάδελφοι, ε, πρόσφατα πριν από δύο μήνες στην Ολομέλεια αποφασίστηκε μία παράταση της εντολής. Αλλά τώρα στη δική μας ε, γνωμοδότηση ε, την οποία πρέπει να εκπονήσουμε πρόκειται για μια νέα εντολή για ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά την άποψή μου. Η πρόταση είναι η ΕΝΙΖΑ να συνεχίσει το έργο της ε, για πέντε χρόνια με μια κάπως τροποποιημένη εντολή και χωρίς ε, να αλλάξει η πρικοδότησή της αλλά με αύξηση του προσωπικού κατά τέσσερα άτομα. Όλοι ξέρουμε ότι όποτε, όταν μιλάμε για τις υπηρεσίες και για το νόημα ε, ή για το παράλογο της επιλογής της έδρας των υπηρεσιών, πάντοτε χρησιμοποιούμε την Ενίζα σαν παράδειγμα προς αποτροπή. Γιατί με το Ηράκλειο που πραγματικά είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτο έχουμε ένα δείγμα για το πώς ε, η έδρα μιας τέτοιας υπηρεσίας ε, δεν μπορεί να ορίζεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όταν προσκαλούνται επιστήμονες να συνεργαστούν με την ΕΝΙΖΑ ή για την ΕΝΙΖΑ ε, και χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα εργασίας για να φτάσουν και για να φύγουν από αυτό το μέρος, δεν είναι ε, ε, εφικτό κάτι τέτοιο. Και η ε, Ενίζα τώρα θα ανοίξει ένα παράρτημα στην Αθήνα τουλάχιστον για κάποιες διεθνείς σκέψεις ή συνέδρια και η χώρα έδρα είναι σύμφωνη. Αλλά τίθεται το θέμα, γύρεται το θέμα κατά πόσο όταν μιλούμε για την Ενίζα ε, και μια παράταση της εντολής της, ε, ή μιλούμε για μια νέα νομική βάση, εάν δεν θα έπρεπε ταυτόχρονα να επιμείνουμε να διευκρινιστεί επιτέλους και το ζήτημα της έδρας και μάλιστα με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε γίνει στο παρελθόν αλλά αυτό δεν χρειάζεται να αναφέρεται ρητά στη δική μας έκθεση, απλώς εγώ το ανέφερα γιατί φυσικά στην Ήτρε ο εισηγητής, ο Charles Chichester, είναι κάποιος ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασχολείται εντατικά με το ζήτημα των υπηρεσιών και αναφέρθηκε στο θέμα αυτό στην έκθεσή του. Εμείς ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε μόνο τις πτυχές του προπολογισμού και αυτές ε, αναφέρονται στο δικό μου σχέδιο, στη δική, μου πρόταση. Κάποιες ε, τροπολογίες που είναι σημαντικές από την άποψη του προπολογισμού. Αλλά έχω εγώ από τη δική μου πλευρά ένα ερώτημα προς την Επιτροπή. Εάν δούμε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι 3,5 άτομα στην υπηρεσία της Επιτροπής θα πρέπει να εργάζονται για να συνεργάζονται για την ενίζα και αυτό στοιχίζει μισό εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, διαρωτώ τι κάνει το αυτή τη στιγμή η Επιτροπή. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αρκεί ένα μόνο πρόσωπο, εάν δεν απατώμε. Και διερωτώ με, είναι απολύτως αναγκαίο στην πράξη να υπάρξουν τρισήμιση μέλη της Επιτροπής που να ασχολούνται με το ΕΝΙΖΑ. Τι θα κάνουν αυτοί. Ε, δεν μπορώ να θέσω το ερώτημα αυτό γιατί ε, πράγματι εδώ πρόκειται για ένα ζήτημα προπολογισμού. Ε, δεν μπορώ να το λύσω με τη νομική βάση, μέσω της νομικής βάσης που προβλέπεται εδώ για την ΕΝΙΖΑ. Θα ήθελα να μου δοθεί μια απάντηση, παρακαλώ. Κατά τα λοιπά, όλα όσα αναφέρουμε και που εμπίπτει στα όρια της αρμοδιότητάς μας επί του προπολογισμού δεν είναι ιδιαίτερος αξιοσημείωτο εδώ ή δεν χρήζει περαιτέρω συζήτηση, γιατί όλοι είμαστε σύμφωνοι. Γιατί πρόκειται, όλο, πρόκειται εδώ για θέματα οποία έχουν συμφωνηθεί ήδη στην ε, διοργανική ομάδα εργασίας ε, μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Και βεβαίως εδώ συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά και όπως είπα δεν χρήζουν περαιτέρω συζήτηση. Δεν εμφανίζουν τις δυσκολίες ή ερωτηματικά. Λοιπόν, αυτά με την Ενίζα και την Έμζα. Αυτά με την Ενίζα, συγγνώμη. Με την Έμζα η κατάσταση διαμορφώνεται κάπως αλλιώς. Γιατί εδώ το θέμα είναι το πώς θα διευρυνθούν οι αρμοδιότητες της Έμζα και ίσως ε, ε, αφού τεθούν τα ερωτήματα προς την Κομισιόν να μας απαντήσει. Αν Γέννησεν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την προσέγγιση που έχετε κι εσείς περιγράψει και τις ε, τροπολογίες που έχετε υποβάλει για τη διαχείριση και άλλα ζητήματα. Είναι θέματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει στην ομάδα εργασία τη διαθεσμική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς. Όμως έχω μια ερώτηση για την ΕΝΙΖΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Υπάρχει ένα στοιχείο που δεν είναι σαφές για την έδρα και για, το, για την έδρα συγκεκριμένα του οργανισμού. Και εδώ φαίνεται να, υπάρχει και, να υπάρχουν και υπηρεσίες αμοιβόμενες για ιδιώτες. Αυτό έχει όντως ε, αρχίσει να λειτουργεί. Μπορεί ο οργανισμός αυτός, η ΕΝΙΖΑ, να κερδίσει χρήματα. Άρα να αυτοχρηματοδοτείται τρόπον την. Yeah. Ευχαριστώ. Να σας πω καταρχάς ότι συμφωνώ πλήρως με τις τροπολογίες σας. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, να δούμε την ενίσχυση στο ευρύτερο πλαίσιο. Το τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός αυτός. Υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊκός οργανισμός για να αυξηθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έχει υποτιμηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα δυναμικός οτιδήποτε και να κάνουμε στον τομέα αυτό δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις. Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια συζητήσεων, αντιπαράθεσης απόψεων, κάποια στιγμή τον, περσινό, τον προηγούμενο μήνα άκουσα τον Επίτροπο να λέει ότι θα εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια στρατηγική για τον κυβερνοχώρο. Αυτή την περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επίσης, το ζήτημα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου αποτελεί τις διμερείς σχέσεις αποτελεί το σημαντικότερο θέμα στις μερείς σχέσεις και μερή συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω δεν θα χρειαστούν δύο ακόμα χρόνια για να εκπονηθεί η στρατηγική αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει την εργασία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και στη συνέχεια μόνο να δούμε ποιο θα είναι ο ρόλος της ε, ΕΝΙΣΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τις εξελίξεις. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πρόκειται για έναν τομεακό οργανισμό και καταλαβαίνετε ότι στον κυβερνοχώρο, στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου χρειάζεται μια, ένας οριζόντιος συντονισμός όχι μόνο η ΕΝΗΣΑ, αλλά και ολόκληρο το πλαίσιο των άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό θα πρέπει να συντονιστούν περισσότερο. Έχετε σαφώ ε, καταπληκτικού εμπειρογνώμονε ε, στην ΕΝΗΣΑ. Ο διευθυντή είναι ένα πολύ άξιο άνθρωπο. Η εντολή όμω που δίνεται στην ΕΝΗΣΑ, η οποία ανανεώνεται προσωρινά κάθε δύο-τρία χρόνια, δεν ευνοεί το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Ε, πραγματικά εδώ πρόκειται για ένα γενικότερο θέμα ε, και μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ, δεν μπορούμε να το κάνουμε μέσω των ε, τροπολογιών. Θα πρέπει να γίνει στην Ήτρε. Εγώ ήδη έθεσα αυτό το ερώτημα πέντε χρόνια και μετά από τρία χρόνια θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση. Όλοι ξέρουμε πώς είναι η δουλειά μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα την περίοδο των πέντε ετών θεωρώ ιδιαίτερα μικρή για να αξιολογήσουμε αυτή την εργασία. Δεν είναι μια νέα υπηρεσία, ήδη υπάρχει, ειδικοί υπάρχουν, αλλά μετά από τρία χρόνια να γίνει αξιολόγηση και να δούμε ποια ήταν η έκβαση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τι θα γίνει μετά από τα πέντε χρόνια. Θα δοθεί πάλι παράταση ε, είναι λίγο το πόδι. Ίσως από την άλλη ε, θα υπάρξει κάποια, ενδεχομένως θα υπάρξει κάποια αλλαγέννη. Η Νέλη Κράους θέλει να λανσάρει το πρόγραμμα κυβερνοασφάλειας ή όταν το έχει παρουσιάσει. Δεν ξέρω, ε, ξέρετε κάτι σχετικά. Μπορείτε να μας απαντήσετε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να απαντήσω σε μερικά από τα όσα τέθηκαν. Η νέα αποστολή του οργανισμού συνίσταται στο να προσφέρει στήριξη και συμβουλές για, τη ρυθμισ... για τις ρυθμιστικές εξελίξεις και ανάγκες. Αυτό είναι η βασική ερμοδιότητα του οργανισμού, αλλά να ασχολείται και με την ε, επιβολή του νόμου και τις αρχές που λειτουργούν στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά σε σχέση με τις βασικές υπηρεσίες για την έδρα και το τι θα γίνει με την ε, εκπνοή της ρήτρα Sunset. Είπατε, Πρόεδρε, ότι αυτά είναι οριζόντια θέματα που καλό είναι να τα δει κανεί στη διαθεσμική οργανή, ε, ομάδα εργασία για του οργανισμού. Χρειαζόμαστε κοινού κανόνε, όλοι μα, για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Για το δικό σα, τώρα συγκεκριμένο ερώτημα για τα συγκεκριμένα καθήκοντα των εργαζομένων της Επιτροπής που έχουν αναλάβει τις σχέσεις με τον οργανισμό. Πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και της λειτουργίας αυτού του οργανισμού, εφόσον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται στο Συμβουλίο. Και ένα συγκεκριμένο καθήκον από πλευρά της Επιτροπής θα είναι να καταγράψουμε τις αρμοδιότητες αυτές που έχουμε αναθέσει, ώστε να τις γνωστοποιήσουμε και στα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ. Ναι. Ε, ε, ε, υπάρχει κάποιος... Υπάρχει ένας ειδικό της ΕΝΙΖΑ, ο οποίος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω απλώς κάτι στην απάντηση του συναδέλφου μου και να αποσαφηνίσω αυτό το οποίο είπατε για τα 3,5 άτομα. Ποιο είστε παρακαλώ. Sorry about that. My name is... Roger από την DG Information Society, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας Πληροφορίας και Desk Officer για την ENISA. Αυτή είναι η θέση μου. Όπως και για άλλους οργανισμούς προβλέπεται ένας Desk Officer και για την ENISA. Αυτό που είπατε για τα 3,5 άτομα ουσιαστικά αφορά όλα τα υπόλοιπα άτομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΝΗΣΑ. Πρόκειται για πάνω από 2,5 άτομα. Αναφερόμαστε σε πολύ περισσότερους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στενή συνεργασία με την ΕΝΗΣΑ το ζήτημα της ασφαλείας των δικτύων, των ασφάλειας των πληροφοριών, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να γίνουν έντονες συζητήσεις. Επομένως, όντως τέτοιες συζητήσεις λαμβάνουν χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και μια πολύ καλή επίβλεψη του έργου της ΕΝΗΣΑ κάθε φορά που καταρτίζουμε το ε, πρόγραμμα εργασίας της. Γίνεται μία συζήτηση στα workshops τα οποία διοργανώνονται σε επιμέρους ομάδες εργασίας και ασχολούμαστε με όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την δημοσιονομική παρακολούθηση, εποπτεία της, του οργανισμού αυτού και το έργο αυτό έχουν αναλάβει αυτά τα 3,5 άτομα. Äh, Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς το ΕΛΚ παρακολουθεί εκ του σύναγκης το ζήτημα αυτό. Καταλαβαίνω πλήρως λοιπόν αυτούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σκεπτικιστές απέναντι στους διαφορετικούς αυτούς οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκύπτουν πολύ περισσότερα ερωτήματα από ότι απαντήσεις πολλές φορές. Ähm, ähm, äh, ναι, η Ενίζα δεν είναι το άψογο παράδειγμα, για να το πω έτσι. Ε, ε, εξαίρετη εργασία επιτελεί μεν. Αυτό είναι το θλιβερό, αλλά δυστυχώς οι συνθήκες που επικρατούν δεν είναι οι καλύτερες. παρόλα αυτά Καταλαβαίνω τι λέτε. Ε, ας πάμε τώρα στην ΕΜΖΑ. Η ΕΜΖΑ είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Και ε, μέσω της συζήτησης που έγινε στην Επιτροπή Μεταφορών ε, τώρα θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες. Γι' αυτό θα αλλάξει ο βασικός κανονισμός για την ΕΜΖΑ και θα πρέπει και εμείς να δώσουμε εδώ σχετικά τη δική μας ε, γνώμη. Ε, εγώ όπως είπα και για την ΕΝΙΖΑ ε, πρόκειται για τις τροπολογίες που ήδη κατέθεσα που αφορούν στον προϋπολογισμό. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να γνωρίζω κατεπηγόντως από την Επιτροπή είναι το εξή. Ήδη ρώτησα την Επιτροπή Μεταφορών και ρώτησα την ίδια την ΕΜΖΑ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έλαβα καμία απάντηση. Η πρόταση της Επιτροπής είναι έξι μέλη του προσωπικού. Nun wissen wir aber selber immer alle, Äh, να αποσπαστούν για, για το νέο τους έργο, για το νέο τους καθήκοντα. Αλλά όλοι γνωρίζομαι, όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές, ότι έχουν ένα περιορισμένο προσωπικό. Πώς μπορεί να εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως σας είπα η Επιτροπή Μεταφορών δεν μπόρεσε να μου δώσει κάποια ικανοποιητική απάντηση. Ε, ελέγχθη μόνο ότι θα γίνουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Ίσως έχετε εσείς μια καλύτερη ιδέα για το πώς αυτοί οι έξι άνθρωποι θα βρεθούν από το redeployment γιατί δεν υπάρχουν, δεν διατίθενται αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάπου εδώ γύρω και περιμένουν θα πρέπει να βρεθούν Πού θα τους βρούμε λοιπόν Thank you, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε η απάντηση θα είναι σύντομη. Είναι ευθύνη των διευθυντών των ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού. Όπως και άλλοι φορές και οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήθηκε από τον οργανισμό να κάνει τη βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων που διατίθενται των ανθρωπίνων συγκεκριμένα πόρων. Η απόσπαση είναι κάτι που η Επιτροπή το πράττει εδώ και χρόνια. Φαίνεται και από τον προπολογισμό του 2012. Και σε άλλους οργανισμούς είχαμε αποσπάσεις και αναδιοργάνωση κάποιες φορές τέθηκαν συγκεκριμένε υποχρεώσει σε κάθε οργανισμό και χρειάστηκε να ανταποκριθεί σε αυτέ τι απαιτήσει. Οπότε κάτι ανάλογο θα, δίνει, θα γίνει και εδώ. Ευχαριστώ. Er Μέχρι τώρα δεν ήταν σε θέση να το κάνει. Κύριε Ρικέ, έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα, για να σας πω μόνο ότι την πρόταση αυτή απόσπασης θα πρέπει να τη δούμε στο πλαίσιο των μελλοντικών δραστηριοτήτων του οργανισμού γιατί θα έχουμε αύξηση των αποστολών του οργανισμού αυτού όσον αφορά τον έλεγχο. Θα γίνει λοιπόν μια επανατοποθέτηση του προσωπικού και θα πρέπει βέβαια αυτή να ανταποκρίνεται στην αύξηση των αποστολών ελέγχου που θα έχει στο μέλλον η ΕΜΣΑ. Στην πράξη ουσιαστικά βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασία η οποία θα αποδειχθεί στο μέλλον πολύ πιο σημαντική. Θα γίνει μια επαντοποθέτηση, μια απόσπαση προσωπικού μικρή στην αρχή, αλλά θα είναι πολύ πιο σημαντική στο μέλλον. Να πω και κάτι ακόμα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους αυτούς που επιτίθενται στους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι τεχνικές υπηρεσίες τελικά, οι οποίες ε, εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να τους καταλογίσουμε τόσο, αρνητικά στοιχεία. Ναι, ε, δεν μπορώ να παρά να συμφωνήσω. Είμαι απολύτω πεπισμένη για κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει να προσθέσω ότι έχουμε πάντοτε υπηρεσίε όταν η ίδια η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει η ίδια, να παράσχει η ίδια τις υπηρεσίες για τις οποίες προβλέπονται αυτές οι υπηρεσίες. Ε, αυτό γίνεται σε κάθε αξιολόγηση όταν θέλει να προβεί στη σύσταση μιας υπηρεσίας και αν το κοιτάξουμε θα δούμε ότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Το θέμα είναι το πώς τελικά μεταχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις υπηρεσίες. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι όλα αυτά είναι εντελώς περιτά, αλλά καμιά φορά στερούνται λογικής. Έχουμε το αίτημα του κυρίου Λεβαντόφσκι για μηδενική αύξηση το επόμενο χρόνο όσον αφορά το προσωπικό. Αλλά τι σημαίνει αυτό μηδενική αύξηση για τις κανονικές ε, θέσεις. Ε, έργου, θα ανθέσουμε το έργο σε άλλες υπηρεσίες. Δεν ξέρω. Ε, αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να την κάνουμε στις 9 Μαΐου με τον αρμόδιο Επίτροπο. Το ζήτημα είναι ε, τι γίνεται με μια τέτοια ιστορία απόσπασης ή αναδιοργάνωσης. Οι θέσει είναι τρεις. Βλέπουμε το σχέδιο προεπλογισμού για αυτό το χρόνο. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά αγνοεί τα δικά μας αιτήματα. Για παράδειγμα, να μην αφαιρέσει τα assigned revenues από τις ε, υπηρεσίες αυτές. Από την άλλη θα πρέπει να πω ότι δεν είστε διατεθειμένοι να προχωρήσετε σε διορθωτικό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή αυτή από το 2004 φρόντισε οι υπηρεσίε κατά τη διάρκεια ε, μιας περίοδου του προϋπολογισμού να να τους δοθεί επιπλέον προσωπικό. Πάντοτε είπαμε ότι αν θέλετε αύξηση του προσωπικού, ε, παρακαλώ να το κάνετε σωστά. Να γίνει αυτό μέσα του προπολογισμού. Μέχρι σήμερα υπάρχουν σχετικά παράπονα. Παρόλο που αυτό δεν είναι σημαντικό για το δικό μας προπολογισμό γιατί θα μπορούσαν να το χρηματοδοτήσουν και οι ίδιοι με τα δικά τους έσοδα. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ε, κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, δική μας ε, στάση. Ίσως δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την σωστή διαδικασία του προπολογισμού, αλλά να λειτουργήσουμε κι εμείς πιο άναρχα. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε λοιπόν ποια είναι, πώς διαφαίνονται οι εξελίξεις. Λοιπόν, 16 ε, Πέμπτου είναι η προθεσμία κατάθεση των τροπολογιών για τις δύο γνωμοδοτήσεις και τον Ιούνιο, στις 15 Ιουνίου, ε, θα πρέπει να ψηφιστούν οι γνωμοδοτήσεις. Μέχρι τις 16 Πέμπτου λοιπόν είναι η προθεσμία. Το Μέχρι το μεσημέρι στις 12 είναι η προθεσμία λήξη για την κατάθεση των τροπολογιών. Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι θα συναντηθούμε πάλι την Πέμπτη. Γεια σας και καλό βράδυ. Α, είσαι καλά, θα πας στο Παλέρμο, ναι, μας το είπες. Ωραία. Ah, das ist am, am, am, das ist am Mittwoch, Agentur. Ah, da bist du auch schon weg. Ja, okay. Ja.